Bene, Καλώς θα ξεκινήσουμε την δημόσια αυτή ακρόαση για ένα θέμα πολύ σημαντικό, το θέμα των δυνατοτήτων της πληροφορικής. θα ήθελα να σας δώσω και κάποιες ε, πληροφορίες για το πώς θα προχωρήσουν οι εργασίες σήμερα. Έχουμε μέχρι τις 5.30 χρόνο. Η Πιλάρντε Καστίγιο θα ξεκινήσει τις ε, παρουσιάσεις, η οποία είναι η συγγήτρια της Επιτροπής Ήτρε. Μετά για 15 λεπτά θα ακούσουμε τους εισηγητές μας. Πέντε εισηγητές. Και στο τέλος κάθε ομιλίας θα έχουμε πέντε λεπτά για κάποια μικρή συζήτηση. Θα δώσω το λόγο στην Πιλάρ πρώτα όμως. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι. Είναι μεγάλη χαρά που κάνουμε αυτή τη συζήτηση για το cloud computing. Θα ήθελα να πω ότι οι δύο άλλοι εισηγητές από άλλες επιτροπές δεν μπορούν να είναι μαζί μας σήμερα. Οπότε δεν θα μπορέσουν να πάρουν το λόγο και να κάνουν παρατηρήσεις. Ίσως αυτό μας αφήνει λίγο χρόνο περισσότερο. Είναι σαφές ότι οι οικονομικές προοπτικές και οι τεχνολογικές προοπτικές του νέφους είναι μεγάλες. Πρόκειται για μια καλή επιχειρηματική ευκαιρία. Αυτό σημαίνει ότι είτε με την παρέμβαση της Ευρώπης είτε χωρίς την παρέμβαση της Ευρώπης το νέφος θα συνεχίσει να αναπτύσσεται αλλά για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες ε, του ψηφιακού νέφους, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάποιες προκλήσεις, έτσι ώστε να ε, έχουμε ένα καλό περιβάλλον για την ανάπτυξή του. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας στα μη τεχνικά θέματα, όπως τα θέματα τα νομικά, ασφάλεια, των δεδομένων, πειρατεία των δεδομένων. Είναι θέματα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η φύση του νέφους προσθέτει θα έλεγα ένα επίπεδο ανασφάλειας σε σχέση με την ασφάλεια της προστασίας των δεδομένων. Δεύτερον, Τελικά οι χρήστες θα πρέπει να είναι σε θέση να ε, έρχονται σε επαφή με τον παροχέα των υπηρεσιών μέσω νέφους με ασφαλή τρόπο. Πρέπει να υπάρχει διαδραστική δυνατότητα επικοινωνίας. Αυτό θα βοηθήσει τον ανταγωνισμό και πολλαπλές παρουσίες νεφών διαθεσίμων και γι' αυτό θα πρέπει να περάσουμε και σε επίπεδα καθορισμού των τεχνολογικών προτύπων. Όχι μόνο λοιπόν λόγω των κερδών σε επίπεδο παραγωγικότητας, αλλά και για λόγους διευκόλυνσης οι πολίτες θα είναι σε θέση να έχουν στη διάθεσή τους ένα καινοτόμο τρόπο επεξεργασίας και μεταφοράς δεδομένων. η δημόσια διοίκηση σαν παράδειγμα θα πρέπει να περάσει πλήρως την ψηφιακή μορφή διάθεσης των υπηρεσιών της. Αυτό είναι βασικό, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει ε, θα έλεγα να χαρακτηρίσει το σύνολο των προσπαθειών που γίνονται στον τομέα της πληροφορικής στην Ευρώπη Θα πρέπει λοιπόν να περάσουν τα κράτη και οι δημόσιες διοικήσεις τους στον ψηφιακό κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω έχει δώσει μια καλή στρατηγική γραμμή στο Κοινοβούλιο και νομίζω ότι εμείς εδώ καλούμεθα να προχωρήσουμε σε κάποιες πιο α, περισσότερες λεπτομέρειες. Καταρχάς θα ήθελα να υπογραμμίσω τη σύνδεση ανάμεσα στην επιδίωξη της βελτίωσης της στρατηγικής για το ψηφιακό νέφος και στην ολοκλήρωση της ψηφιακής αγοράς. Το νέφος υπογραμμίζει την ανάγκη για εναρμόνιση και μπορεί να λειτουργήσει επιταχυντικά για την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Έχουμε ένα εξαιρετικό πάνελ εδώ το οποίο θα αντιμετωπίσει τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ε, το νέφος. Η κατάσταση της αγοράς, τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν ε, οι δημόσιες υπηρεσίες όταν περνούν στο νέφος, τα επίπεδα τα οποία πρέπει να είναι τεχνολογικά ε, έγκυρα, και πρέπει να δούμε επίσης και την αντίληψη του κοινού για τη στρατηγική των νεφών. Όπως ξέρετε η κυρία Σαρτζεντίνη και μία άλλη συγγήτρια δεν μπορεί να είναι μαζί μας σήμερα, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε με τον πρώτο ομιλητή, τον κύριο Στέφανο Μπράτα. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί βουλευτές, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσω τις απόψεις της τηλεφώνικα για τη συζήτηση για τον ΕΦΟΣ. Είμαι ο Στέφανο Φράτα, δουλεύω για την τηλεφώνικα Digital, η οποία είναι θηγατρική της τηλεφωνικά που αναπτύσσει όλα τα νέα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο. Και είμαστε αναμειγμένοι και στην συζήτηση αλλά και στη βιομηχανία που αφορά το νέφο. Χαίρομαι λοιπόν που βρίσκομαι εδώ σήμερα για να μοιραστώ μαζί σα κάποιε ιδέε για το νέφο. Καταρχά, το πρώτο που θα ήθελα σήμερα να τονίσω είναι να αναφερθώ σε κάποιε παρανοήσει που υπάρχουν σε ό,τι αφορά το νέφο και το τι σημαίνει για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Προτού ξεκινήσουμε να μιλάμε για τις ε, αντιλήψεις αυτές που επικρατούν, τις λανθασμένες συχνά αντιλήψεις, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι αν και σήμερα μιλάμε πάρα πολύ για το cloud, το νέφος και το τι ακριβώς είναι, η αλήθεια είναι ότι οι εξαποστάσεις υπηρεσίες ήταν μαζί μας από την αρχή, από την επαρχή του διαδικτύου. Αν θυμηθείτε το πρώτο ε, email που είχατε, τον πρώτο λογαριασμό email πριν από 20 χρόνια, ήταν είτε Hotmail, είτε Yahoo, είτε Altavista, και αυτό, αν θέλετε, είναι μια υπηρεσία νέφους, πριν από 20 χρόνια ήδη. Και τα online ε, ημερολόγια, ε, ατζέντε ήταν όλα τέτοιε υπηρεσίε εξ αποστάσεως. Άρα από αυτήν την άποψη τι άλλαξε πρόσφατα τα τελευταία χρόνια. Τι μας ε, έκανε να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση για το νέφος. Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία συνέβαλαν σαφώ στις πρόσφατε εξελίξει. Καταρχάς, η τεράστια αύξηση στον χώρο των αποθηκευτικών σε πιο χαμηλές τιμές. Ε, ο όγκος των δεδομένων που μπορούμε σήμερα να αποθηκεύσουμε δεν συγκρίνεται με αυτά που μπορούσαμε να αποθηκεύσουμε πριν από κάποια χρόνια. Κατά δεύτερον, η βελτίωση της ποιότητας και της ταχύτητας που παρέχουν οι πάροχοι, τα δίκτυα για να έχουμε πιο γρήγορο δίκτυο για τον καταναλωτή, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλέον και για να, ανεβαστεί, να ανεβάσουμε πιο πολύ υλικό. Το τρίτο είναι ασφαλώς η ανάπτυξη νέων συσκευών, όπως τα smartphone, τα tablet, όλοι σας ε, με τα iPhone μπορείτε να ανεβάσετε τη μουσική σας στο iCloud και με άλλες συσκευές ασφαλώς και ασφαλώς η γενικότερη αποδοχή της κουλτούρας του διαδικτύου. Όλοι αυτοί οι παράγοντες λοιπόν ήταν παρόντες τα τελευταία χρόνια και δημιούργησαν αυτό το περιβάλλον του νεφού στο οποίο σήμερα συζητάμε. Ωστόσο, μπορούμε να πούμε ότι κάθε ένας από αυτούς τους παράγοντες υποστηρίζει ένα διαφορετικό επιχειρηματικό μοντέλο για τα smartphones. Τι σημαίνουν εκατομμύρια άνθρωποι μπορούν να ανεβάσουν μικρές ποσότητες, μικρό όγκο δεδομένων στο δίκτυο. Και εκ παραλλήλου η μεγάλη ταχύτητα σημαίνει ότι οι μεγάλοι όμιλοι δεν χρειάζονται να αποθηκεύουν τοπικά πλέον τα στοιχεία τους, τα δεδομένα τους. Μπορούν να έχουν υπηρεσίες βάσει του νέφους και έτσι να έχουν πρόσβαση από όλες τις θηγατρικές του ομίλου σε όλο τον κόσμο. Για παράδειγμα, στην τηλεφωνικά digital, για παράδειγμα, πρόσφατα εφαρμόσαμε μια βάση δεδομένων ε, ανθρώπινου δυναμικού αποκλειστικά στο νέφος. Αυτό τι σημαίνει ότι η τηλεφώνικα digital που δουλεύει στη Μαδρίτη, στο Σαο Πάολο, στο Λονδίνο, ε, οπουδήποτε στον κόσμο έχουν όλη πρόσβαση στο ίδιο έγγραφο το οποίο αποθηκεύεται ε, στο νέφος. Από που και αν βρίσκεται κανείς, μέσω του τάμπλετ του έχει έτσι πρόσβαση στο ίδιο έγγραφο. Βλέποντας λοιπόν τα διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία υποστηρίζει η αρχή του νέφους, μπορεί κανείς να συμφωνήσει με αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν λέει ότι είναι πάρα πολύ χαλαρός ο ορισμός του νέφους. Όντως είναι πολύ χαλαρός ο ορισμός. Να μην το ξεχνάμε αυτό όταν μιλάμε για οποιοδήποτε μελλοντική ενδεχόμενη νομοθεσία που θα επηρεάσει τον νέφους. Θα ήθελα να ξεκινήσω να κοιτάμε, να σας αναφερθώ σε κάποιες από τις παραμείσεις λοιπόν, που επικρατούν για τον νέφος. Η πρώτη είναι η εξής ότι το νέφος εγγυάται καλύτερη προστασία των δεδομένων. Η μετάβαση σε μια βιομηχανία εξ αποστάσεως, αν θέλετε, μέσω του νέφους, θα είναι πιο ασφαλής από τη τρέχουσα κατάσταση. Τι γίνεται με τις μικρές επιχειρήσεις αποθηκεύουν στο σκληρό τους δίσκο, σε ένα σερβερ που έχουν ίσως στην αποθήκη τους, ε, τα δεδομένα. Αν πιστεύουμε απαραίτητα ότι αυτές οι εταιρείε ε, εφαρμόζουν ε, πρότυπα υψηλή ασφάλειας, είναι σχετικό. Ξέρουμε πόσα δεδομένα χάνονται καθημερινά στην Ευρώπη, επειδή είναι πολύ χαμηλά τα πρότυπα προστασία των δεδομένων. Επειδή, για παράδειγμα, έχει πλημμυρίσει ένα υπόγειο, χάνονται αυτά λοιπόν τα δεδομένα ε, χάνονται για παράδειγμα επειδή μπορεί να χαλάσει ο υπολογιστή, επειδή χρησιμοποιεί μια παροχημένη έκδοση των Windows και έτσι ε, σε πολλές περιπτώσεις χάνεται η πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία όταν είναι αποθηκευμένα σε ένα σκληρό σε ένα σερβερ. Εκ παραλλήλου πιστεύουμε ότι η μέση επιχείρηση, η μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί πραγματικά να επενδύσει για να έχει, για παράδειγμα, προστασία στο ασύρματο δίκτυό τους. Ξέρουμε τι θα συμβεί όταν οι μικρές επιχειρήσεις ή οι μικροί επαγγελματίες φέρνουν τα λάπτο τους και τα πηγαίνουν στο κατάστημα της γειτονιάς για επισκευή. Ξέρουμε ποιος έχει πρόσβαση στο υλικό αυτό. Ξέρουμε τι ε, μέτρα ασφαλείας εφαρμόζονται. Αυτό δεν το ξέρουμε. Ενώ το νέφος ε, συμβάλλει στην ασφάλεια των δεδομένων αυτών. Γιατί εμείς ως πάροχοι του νέφους ε, δουλεύουμε σε θέματα ασφάλειας. Η πρόσβαση εξ αποστάσεως που παρέχουν οι μεγάλοι παροχοί νεφούς αποτελούν λοιπόν αποτελεί μια σημαντική βελτίωση για την προστασία των δεδομένων. Να μην θεωρήσουμε ότι αυτή η μετάβαση από το τοπικό επίπεδο στο κεντρικό επίπεδο για την αποθήκευση των δεδομένων σημαίνει απαραίτητα χαμηλότερη ασφάλεια. Υπάρχουν κίνδυνοι και στο τοπικό επίπεδο. Σκεφτείτε λοιπόν αυτή την προσέγγιση και σκεφτείτε και να έχουμε υπόψη αυτή την προσέγγιση σε ό,τι αφορά οποιαδήποτε κατάρτιση νομοθεσία που θα αφορά το νέφο. Ε, είναι αρκετά απλό να καταλάβει κανείς γιατί η τηλεφωνικά θέλει να ε, αρθούν τα εμπόδια για την ανάπτυξη του νέφους ε, στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Θα πρέπει να προάγουμε μια τέτοια πρόταση ε, για την πρόθεση του νέφους, για να προωθήσουμε την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κλάδου και όλης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας από τους ε, επαγγελματίες, από τους μικρούς επαγγελματίες μέχρι τις μεγάλες πολυεθνικές. Αλλά για να πετύχει η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να έρθουν κάποια από τα σημερινά και μελλοντικά εμπόδια που θα μπορούσαν να εμποδίσουν τη μελλοντική ανάπτυξη του νεφους. Και όπως είπε η κυρία Δελκαστή, το πιο σημαντικό πράγμα εδώ είναι ότι εδώ είμαστε για να ενισχύσουμε την ενιαία αγορά και το νέφος μπορεί να συνδράμει προς την κατεύθυνση αυτή. Αλλά για να πετύχουμε μια ενιαία ψηφιακή αγορά θα πρέπει να καταργήσουμε κάποια από τα εμπόδια τα οποία υφίστανται σήμερα και τα οποία υφίστανται σε διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες αλλά επηρεάζουν και τον έφος. Λίγα λεπτά λοιπόν θα ήθελα να αφιερώσω για να ε, σας πω ποια είναι τα εμπόδια αυτό. Καταρχάς, χρειαζόμαστε μια ενιαία ε, μια ενιαία, αν θέλετε, ενιαίους κανόνες για την ιδιωτική σφαίρα που θα ισχύει σε όλο τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι παραγραμματικά κρίσιμη σημασία για να πετύχουν οι υπηρεσίες νέφους ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για πολλές άλλες υπηρεσίες βέβαια ιδιαίτερα για τις υπηρεσίες εκείνες που συναγωνίζονται μεγάλες αμερικάνικες εταιρείε που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες και ε, σε άλλες χώρες εκτός της Ένωσης. Χρειαζόμαστε οικονομίες κλίμακας ε, στο νέφος για να μπορούμε να έχουμε επενδύσεις σε ένα προϊόν από όσο το δυνατόν πιο πολλά άτομα γίνεται, ιδιαίτερα όπως σας είπα για να συναγωνιστούμε τους άλλους παρόχους. Σήμερα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Σήμερα έχουμε μόνο εθνικές αγορές, γιατί κάθε κράτος μέλος έχει διαφορετικές νομικές προδιαγραφές. Αυτό το διαπιστώνουμε πολύ συχνά στην τηλεφωνικά digital, όπως ε, προσπαθούμε να αναπτύξουμε ένα προϊόν και βλέπουμε ε, πώς πωλείται αυτό το προϊόν στις διάφορες χώρες που δραστηριοποιείται η τηλεφώνικα digital και συχνά είναι δύσκολα τα πράγματα γιατί υπάρχουν διάφοροι παράγοντες διαφορετικοί από χώρα σε χώρα σε ό,τι αφορά την προστασία των ε, καταναλωτών, τα θέματα ιδιωτικής σφαίρας, τα θέματα τα φορολογικά. Όλα αυτά τα εμπόδια θα πρέπει να αρθούν, να εναρμονιστούν ε, οι αγορέ προκειμένου να υπάρχει όντω μια ενιαία αγορά για τι ψηφιακέ υπηρεσίε και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τι υπηρεσίε του νεφού. Για να δημιουργηθεί λοιπόν μια πραγματική αγορά ενιαία για, τα ψηφια για τις ψηφιακές υπηρεσίες και για να φτάσουμε σε ένα ε, χωρίς προηγούμενο επίπεδο ε, παροχής υπηρεσιών. Ωστόσο, δεν ε, χρειαζόμαστε μία συγκεκριμένη, αν θέλετε, ομάδα κανόνων για την ιδιωτική σφαίρα σε ό,τι αφορά τον έφο Το νέφος δεν είναι πιο επικίνδυνο απαραίτητα από τη σημερινή κατάσταση. Δεν υπάρχει κανένας λόγος γιατί ο για... για τους οποίους η νέα νομοθεσία για την ιδιωτική σφαίρα θα πρέπει να αυξήσει την ευθύνη και τις περιορισμούς στον έφο. Θεωρούμε ότι όλες οι δραστηριότητες που υπάρχουν στον έφο είναι εισάξεις με τι σημερινέ ε, δραστηριότητε. Και γι' αυτό η διαχωρισμό μεταξύ της επεξεργασίας των δεδομένων ήταν πάντα ένα βασικό στοιχείο στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και με πολύ, ε, πολύ καρποφόρο μέσο που ήταν πολύ χρήσιμο για την ε, διεργασία και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Δεν βλέπουμε γιατί θα πρέπει να υπάρξει κάτι διαφορετικό ως πρόβλεψη για τον έφος. Τρίτο σημείο, θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι μπορεί η γεωγραφική ομογένεια να είναι κάτι βασικό. Χρειαζόμαστε λοιπόν του ίδιου κανόνε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο πράγμα η ομογένεια των ε, προϊόντων. Υπάρχουν διάφοροι κίνδυνοι σε ό,τι αφορά την ιδιωτική σφαίρα και την ασφάλεια, σε ό,τι αφορά κάθε ξεχωριστή δραστηριότητα στο νεφο. Είναι πολύ τρογενεί λοιπόν αυτέ οι υπηρεσίε και ο μοναδικό κοινό παράγοντα είναι η εξαποστάσεω πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή οποιαδήποτε κανόνα που θα ίσχυε σε υπηρεσίες ε, για τον ε, φως, είτε πρόκειται για ασφάλεια, προστασία καταναλωτή, γενική όρεκη. Θα πρέπει να επιδεικνύει την απαραίτητη ευελιξία προκειμένου για να ισχύει σε όλες τις υπηρεσίε του νεφού. Κατά τέταρτον, θα πρέπει να αποφύγουμε επιβολή προτύπων και ειδικών ε, ορίων ποιότητας σε αυτό το μη ομογενές, αν θέλετε, τοπίο καλωσορίζουμε ασφαλώς ε, κάποια συγκεκριμένα όρια, αλλά και πάλι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το νεφο είναι κάτι το πολύ ευρύ, που περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές υπηρεσίες και προϊόντα. Και αυτά που ισχύουν για το ένα προϊόν μπορεί να μην ισχύουν και για κάποιο άλλο. Η τηλεφώνικα αποτελεί ένα βασικό φορέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η εμπειρία μα μας καταδεικνύει ότι τα τεχνικά πρότυπα και τα πρότυπα ποιότητα σε, σε ό,τι αφορά τον έφο, που επιβάλλονται για παράδειγμα από μια τράπεζα δεν είναι ανάγκη να συνάδουν με τις ε, ανάγκες για παράδειγμα του καταναλωτή που θέλει να κατεβάσει κάτι στο iPhone ή του για παράδειγμα μικρού φούρναρη της γωνίας που χρησιμοποιεί τον έφος. Δεν χρειάζεται λοιπόν να υπάρχουν τα ίδια και για τους ε, όλους τους καταναλωτές. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να μεταφραστούν σε νομοθεσία. Τελευταίο ζήτημα, τα θέματα κινητής ε, φορετότητας. Θεωρώ δεν χρειάζεται να είμαστε πιο πατητικοί σε ό,τι αφορά τη φορητότητα στο νέφος από ότι ε, στον κόσμο offline. Θέλουμε τα συστήματα, για παράδειγμα, θέλουμε να επιβάλλουμε υπερβολική και μάλλον ε, υποχρεωτική σε εφαρμογές ε, λογισμικού. Δεν κάνουμε κάτι τέτοιο. Θα πρέπει λοιπόν η φορητότητα να είναι ένα επιπλέον στοιχείο το οποίο θα ληφθεί υπόψη σε μια, ανταγωνιστική αγορά. Δεν ε, αφορά αυτό όμως κάθε ε, καταναλωτή απαραίτητα και πρέπει ο καταναλωτής να, ξέρει, να μπορεί να, να επιλέξει το που θέλει. Για να ε, κλείσω και να σας παρουσιάσω όλα τα στοιχεία ξανά. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία βασικά τα οποία θα πρέπει να έχουμε υπόψη πριν αρχίσουμε να εξετάσουμε οποιαδήποτε νέα ρύθμιση του νεφούς. Καταρχάς, ότι η οθέτηση ε, τέτοιων υπηρεσιών θα οδηγήσει σε μία βελτίωση σε ό,τι αφορά την ιδιωτική σφαίρα, την προστασία των δεδομένων και την διαθεσιμότητα των δεδομένων. Κατά δεύτερον, ότι είναι καιρό να δείξουμε ευελιξία σε ό,τι αφορά τι βέλτιστε πρακτικέ, τι κατευθυντήριε γραμμέ, τα πρότυπα, κώδικα συμπεριφορά. Θα πρέπει να είμαστε ευέλικτοι, να μην είναι ε, υπερβολικά αυστηρή η σχετική νομοθεσία. Κατά τρίτον, σε ό,τι αφορά τα θέματα ασφάλειας και θετικής σφαίρας προστασίας του καταναλωτή, οποιαδήποτε νομοθεσία θα πρέπει, που θα ισχύει για το νέφος, θα πρέπει να μην ε, χρήζει ειδικών κανόνων και δευθυνήσεων. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ωραία, λοιπόν, έχει ζητήσει το λόγο... Α. Ε, οι ερωτήσεις καλύτερα να γίνουν στο τέλος. Δεν χειριστούμε εύκολο αυτό, καθώς δεν είναι πολλοί κόσμο εδώ. Ευχαριστούμε πολύ για όλη αυτή την πολύ καλά διαρθρωμένη παρουσίαση και όλα αυτά τα μηνύματα. Στη δεύτερη θέση τώρα για τις δημόσιες συμβάσεις και το απολογιστικό νέφος ε, έχω ε, τον Φίλιπ Φαν Ευχαριστώ πολύ. Είμαι ο Φίλιπ Αβερμάτ, ε, Διευθυντή ε, Δημοσίων Συμβάσεων και Υπολογιστικού Νέφου τη Σχετική Γενική Διεύθυνση του Κοινοβουλίου. Και σε αυτή την παρουσίαση θα σας δώσω και πρακτικά παραδείγματα για να σας δείξω ότι δεν είναι μόνο οι θεωρητικές, ε, τα πράγματα δεν είναι μόνο θεωρητικά και δεν είναι μόνο αυτά που πρέπει να μας καθοδηγούν. Τώρα όσον αφορά την ορολογία, το cloud computing είναι μεγάλη προτεραιότητα από πέρυσι. σε κάποιες ε, εταιρείες ονομάζεται hosting, virtualization ως υπηρεσία. Εικονικοποίηση δηλαδή, φιλοξενία πολύ κοινή όρη αυτή συνήθως. Κάποιες προϋποθέσεις. Η μετάβαση στο υπολογιστικό νέφος απαιτεί οριμότητα των επιχειρήσεων και των οργανισμών, όχι μόνο από τεχνική άποψη, που θα Πρέπει να αλλάξει και η εξωτερική συνδεσιμότητα και οι συσκευέ πρόσβαση. Σε ορισμένε μικρομεσαίε επιχειρήσει τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά από τι μεγαλύτερε εταιρείε. Καλή υπάρχουσα λειτουργική υποδομή υποστήριξης είναι απαραίτητη για να συνοδεύει την αλλαγή αλλά και για να αλλάξει το δικό τη ρόλο από την υποστήριξη των εσωτερικών χρηστών στο να γίνει η διασύνδεση μεταξύ χρηστών και των παρόχων υπολογιστικού νέφους. Και φυσικά όταν κάποιος θέλει να οικοδομήσει ένα καλό χάρτη πρέπει να μπορεί να προσαρμόσει τις απαιτήσει του στις υπηρεσίες, τις λειτουργικές απαιτήσει της υπηρεσίας και να μην πιστεύουμε πια ότι όπως το παρελθόν ξεκινάμε σκεπτόμενοι αν χρειάζομαι μια νέα εφαρμογή ή ένα νέο μοντέλο. Είναι καλύτερο να αλλάξουμε νοοτροπία, να χαρτογραφήσουμε τις απαιτήσει μας με βάση τις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίε του υπολογιστικού νέφου. Κατά προτίμηση. Τώρα, πιο σχετικά με τις δημοσίες συμβάσει και τις άμεσες και έμεσε επιπτώσεις του υπολογιστικού νεφού στις δημοσιε συμβάσει, πρώτα απ' όλα έχουμε τον κατακρεματισμό. Θα έχουμε λιγότερες ή περισσότερες συμβάσει να διαχειριστούμε, εάν επιλέξουμε το υπολογιστικό νέφος. Είναι πολύ πιθανότητα για την αγορά υλικού, hardware, θα δούμε σημαντική μείωση των αριθμών συμβάσεων που χρειάζεται κανείς να διαχειρίζεται. Ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό ανατίθεται σε εξωτερικούς συνεργάτες ένα μεγάλο κομμάτι των, ε, του εξοπλισμού και οι αδείες λογισμικού θα μειωθούν σε μεγάλο ποσοστό τα, οι συμβάσεις δικτύων μπορεί να παραμένουν ίδιες, ίσως να χρειαστούν κάποια ενίσχυση ώστε να υπάρξει καλύτερη συνδεσιμότητα. Όσον αφορά τις υπηρεσίες, εκεί μπορεί κάποιος να εξενηθήσει να λειτουργεί, να συνεργάζεται με ένα εσωτερικό ή εξωτερικό ανάδοχο και εφόσον αλλάξει σε υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους μπορεί να έχει να διαχειριστεί περισσότερες συμβάσεις. Επίσης υπάρχει μια έμεση επίπτωση στην ε, επιμελητία, στο logistics. Χρειάζεται κανείς ε, λιγότερα τετραγωνικά μέτρα, λιγότερους χώρους όταν αποθηκεύει τα δεδομένα εκτός της εταιρεία. Και το ερώτημα ε, εκεί είναι πώς συμβάσεις υπολογιστικού νεύους μπορεί να διαχειριστεί ο οργανισμός σας, η εταιρεία σας και χρειάζεται μετάβαση σε μια μεγάλη εταιρεία από τοπικά ε, συμβόλαια νέφους, ενώ σε μια μικρομεσαία επιχείρηση λειτουργούν τα πράγματα σε ένα πολύ μικρό περιβάλλον και υπάρχει ενδεχομένω αλληλεπίδραση εκεί με πολλούς παρόχους υπολογιστικού νέφους. Θα επηρεάσει αυτό και την αξία των συμβασιών σας. Ε, θεωρητικά ναι. Θα έχετε μεγαλύτερες, περισσότερες μάλλον συμβάσεις, συγγνώμη, χαμηλότερης αξίας διότι κατανέμονται οι προσπαθείς και υπηρεσίες που αγοράζει κανείς ε, στο υπολογιστικό νέφος. Επίσης θα επηρεαστούν οι εγγυήσει που θα απαιτείται από τους αναδόχους. Με τη σημερινή κατάσταση στις συμβάσεις απαιτείται συχνά η οικονομική ικανότητα ενός αναδόχου που στο υπολογιστικό νέφος δεν έχει νόημα. Καθώς δεν μπορείτε να γνωρίζετε πού βρίσκεται ο εξοπλισμός και πώς έχει, επηρεάζει τις επιδόσεις της εταιρείας. Ενώ η απέτηση για μια επαγγελματική ασφάλεια, διασφάλιση, αυτό είναι σημαντικό όταν το συμβόλαιο δεν εκτελείται όπως θα θέλατε. Και δεν έχετε καμία επαφή με τον πάροχο γιατί δεν βρίσκεται στο χώρο σας, δεν μπορεί να έρθει στο χώρο σας, δεν έχει εξοπλισμό στο χώρο σας, οπότε δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα εκτός από το να επικαλεστείτε την επαγγελματική ασφάλεια. Πολύ συχνά έχουμε μία μόνο εφαρμόσιμη νομοθεσία στα τρέχοντα συμβόλαια. Τα, τα συμβόλαια υπολογιστικού νέφους είναι λίγο πιο περίπλοκα να κάνει κανείς ε, ε, ε, προσφυγή στη χώρα του πελάτη, του παρόχου ή κάπου αλλού, ενδεχομένως στη χώρα όπου λειτουργούν ή βρίσκονται οι, εξοπλισμοί από που γίνεται η διαχείρισή τους. Ενδεχομένως ο παροχός σας να είναι μια μητρική, μια θηγατρική εταιρεία και τα πράγματα που αφορούν εσάς να εκτελούνται κάπου αλλού. Και εδώ έρχομαι στο επόμενο σημείο της άγνωστης τοποθεσίας. Χρειάζεστε λοιπόν πολύ μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον συνεργάτη σας. Δεν είναι μόνο θέμα ασφάλειας των δεδομένων πληροφορικής, είναι και θέμα φυσικής ασφάλειας. Τι γίνεται σε περίπτωση που οι εγκαταστάσεις του παρόχου βρίσκονται στη βεριτό δεν το γνωρίζετε. Και αυτό μπορεί να αποτελέσει ζήτημα. Και φυσικά όταν τα πράγματα δεν πάνε πολύ καλά, εκεί τίθεται το θέμα της επίλυσης διενέξεων και το ε, δικαστήριο στο οποίο θα προσφύγει κανείς. Το που θα βρίσκεται, σε ποια δικαιοδοσία και κατά πόσο θα υπάρχει κάποια ως μηχανισμός επίλυσης διενέξεων με μεσολάβησης με την κατάλληλη δομή. Ένα άλλο ζήτημα φυσικά είναι το ζήτημα της προστασίας δεδομένων ε, που θα πρέπει να απεικονίζεται κάπως τη συμβάση. Αλλά πώς. Πώς να περιορίσει κανείς να το περιορίσει στις 27 χώρες της Ευρώπης. Ε, όταν έχουμε την τοποθεσία του eBay, του Βελγίου για παράδειγμα και δεν λειτουργεί, μας ανακατευθύνει κανονικά στο αμερικάνικη ιστοσελίδα σελίδα σύνδεσης τα δεδομένα σας λοιπόν πού βρίσκονται. Μια άλλη πτυχή που αφορά την προστασία των δεδομένων πιο δύσκολη για τις συμβάσει κατά την απόψή μου είναι τι γίνεται σε περίπτωση απώλειας των δεδομένων ή σε περίπτωση παράνομης χρήσης τους εθελουσίως ή όχι λόγω παρέμβαση κάποιων hacker ή λόγω κάποιες απώλειας ένα άλλο θέμα αφορά την ιδιοκτησία των δεδομένων, των αποθηκευμένων δεδομένων, διότι είναι δικά σας δεδομένα αρχικά, αλλά δεν ξέρουμε πού θα αποθηκευτούν και εν τέλει κανείς δεν ξέρετε, εσείς δεν ξέρετε κατά πώς θα παραμείνουν δικά σας. Το ίδιο ισχύει για τις αποθηκευμένες διαδικασίες και φόρμες εργασίες. στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει ξεκινήσει ένα τεράστιο πρόγραμμα υλοποίησης μιας ροής εργασιών διανομής ταυτοτήτων. Στο τέλος, δεν ήταν ιδιοκτήτης ούτε της ροής εργασιών ούτε των δεδομένων και χρειάστηκε να πληρώσουν 3 εκατομμύρια λίρες για να επανακτήσουν τα δεδομένα τους και όλες τις διαδικασίες στα δικά τους μηχανήματα και στους χώρους τους. Το επόμενο φυσικά σημείο είναι το ερώτημα του τι γίνεται με τα δεδομένα που παράγονται στο υπολογιστικό νέφος. Παραμένουν δικά σας ή μήπως θα βρείτε ε, ρήτρες σε μικρά γράμματα μέσα στα συμβάσεις που θα λένε ότι το σύστημα χύψη ε, βρίσκεται, ανήκει στην εταιρεία που το παρήγαγε. Επίσης πρέπει να προσέξουμε τη σύνταξη των συμβάσεων όσον αφορά τη μεταφορά δεδομένων στο υπολογιστικό νέφος. Συνήθως αυτό είναι εύκολο η μεταφορά δεδομένων και φυσικά ο πάροχος θα είναι διατεθειμένος να συνεργαστεί μαζί σας, αλλά φυσικά εν τέλει αν δεν έχετε προβλέψει ένα σχέδιο διαχείρισης εξόδου θα καταλήξετε σε μια κατάσταση που θα μπορείτε να ανακτήσετε τα δεδομένα σας ή που θα καταλήξετε σε ατέρμονες, οδυνηρές διαπραγματεύσεις που θα σας κοστίσουν πολύ ακριβά. θα πρέπει να έχει, προτιμάτε συμβάσεις επικεντρωμένες στους πελάτες ώστε να επιλέγετε αυτό που θέλετε εσείς να, όπως κάνετε και με τους ε, φορείς τηλεφωνικών επικοινωνιών. Όταν θέλετε να, επισκευάσετε, να αγοράσετε μια τηλεφωνική γραμμή ή μια τηλεφωνική σύνδεση, πάτε σε έναν πάροχο και αποφασίζετε αν θα την αγοράσετε ή όχι, αλλά δεν αλλάζετε τις ρήτρε. Όταν είστε μια μικρομεσαία επιχείρηση, είναι πολύ πιθανό να γίνει το ίδιο με τους μεγάλους παρόχους υπολογιστικού νεύους. Επίσης υπάρχουν κάποιες πρακτικές πτυχές ότι αν δεν τα φροντίσετε όλα αυτά η υλοποίηση μπορεί να είναι δύσκολη. Η υποστήριξη πελατών επίσης και οι ωραίες ζώνες ε, έχουν σχέση με όλα αυτά. Τις προάλλες ε, είχαμε την εμπειρία υποστήριξη των χρηστών 9 με 5 στη Γαλλία αλλά η έδρα του ήταν στο Λονδίνο, στα αγγλικά. Οπότε ήταν 8 με 4 και η επόμενη λύση είναι ότι πληρώνεται για την υποστήριξη 24 ώρες το 24ωρο, διότι δεν έχει, γίνει, δεν έχει μεσολαβήσει διαπραγμάτευση. και αυτό είναι ένα έμεσο κόστος. Όσον αφορά τις ε, άδειες παροχής υπηρεσίας, επίπεδου υπηρεσίας, το service level agreement, τα SLA όπως λέμε, και αυτό είναι ένα ζήτημα, θα καθοδηγείται από τον πελάτη, από τον πάροχο και κατά πόσο μπορέσει η συμφωνία να είναι εξισορροπημένη. Και τι γίνεται σε περίπτωση βλάβης, διακοπής της υπηρεσίας, η προσωρινή διακοπή της υπηρεσίας, τι γίνεται σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμος ο πάροχος για να λύσει το πρόβλημα. Μπορεί να έχετε άλλες απαιτήσεις ε, ε, για κάποιον συγκεκριμένο τομέα, α πούμε. πώ θα αντισταθμίσετε ε, τα πράγματα σε περίπτωση απώλεια των δεδομένων, απώλεια τη ακαιρεότητα των δεδομένων ή κατάχρηση των δεδομένων και ιδιαίτερα κρίσιμων δεδομένων. Το ίδιο ισχύει και για τις αναφορές ε, βλαβών που η παρακολούθηση μπορεί να μην είναι αντικειμενική. Μπορεί να παρακολουθούνται μόνο το 50%. Και φυσικά όσον αφορά τις αποζημιώσεις και τις ποινές, ποιο επίπεδο έχει δημιουργήσει το πρόβλημα και τι αποδεικτικά στοιχεία έχετε εσείς για να ζητήσετε αποζημίωση. Διότι φυσικά για τον πάροχο του υπολογιστικού νέφους είναι πολύ εύκολο να πει, ξέρετε, ο κόμβος του διαδικτύου στη Σουηδία έχει πρόβλημα. Δεν φταίμε εμείς. Φταίμε αυτοί. Και έχω και ένα πολύ πρακτικό παράδειγμα μια τράπεζα που είχε αναθέσει κάποιες υπηρεσίες στην Ινδία. Ένα μέρος του δικτύου βρισκόταν στην Αίγυπτο και η σύνδεση με την Ινδία δεν ήταν επαρκής και δεν λειτουργούσε αυτή η σύνδεση για τρεις μέρες. Ένα άλλο ζήτημα που χρήζει προσοχής ε, είναι ο έλεγχος του κόστους όταν κανείς έχει τα μηχανήματα στο χώρο του, οι τιμές είναι σταθερές, πολύ ε, συχνά γνωρίζει κανείς τι θα πληρώσει. Συνήθως δεν χρειάζεται μεγάλη επένδυση αρχική στο cloud computing, αλλά συμβαίνει το ίδιο με την τηλεφωνία. Αγοράζετε μια κάρτα για το κινητό σας και δεν έχετε ιδέα πόσο θα κοστίσει Υπάρχει το ίδιο πρόβλημα ελέγχου του κόστου όπως και με το υπολογιστικό νύφος. Αγοράζετε 10 τεραμπάιτα χώρο αποθήκευσης και με ένα-δυο κλικ παίρνετε άλλα δύο, άλλα τρία και εν τέλει το λογαριασμό που σας έρχεται δεν ήταν καθόλου αυτό που περιμένατε στις εκτιμήσεις και βάσει του προπολογισμού σας. Επόμενα όμως ε, είναι λίγα και πιο τεχνικά θέματα και θα τα εξετάσουν οι άλλοι συνάδελφοι. Χρειάζεστε μια εφεδρική λύση. Θα κάνετε κρυπτογράφηση για λόγους ασφαλείας, παρακολούθηση, πώς μπορείτε να παρακολουθείτε τι συμβαίνει. Και φυσικά το υπολογιστικό νέφος δεν είναι η θαυματουργή τεχνολογία, η μόνη θαυματουργή τεχνολογία πρέπει να ληφθεί υπόψη το ενδεχόμενο χρήστη μαζί με άλλες υπάρξεις τεχνολογίες για να Καταλήξουμε λοιπόν εδώ με τα όσα λέει η Κομισιόν. Χρειαζόμαστε ασφαλείς όρους και συνθήκες συμβάσεις φυσικά είναι αναγκαίο. Αλλά πολλά πράγματα πρέπει να ληφθούν υπόψη, πολύ περισσότερα από ότι στις κλασικές συμβάσεις που γνωρίζουμε σήμερα. Είναι αδύνατο να εισάγουμε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις. Πρέπει να έχουμε και τυποποιημένες SLA, Service Level Agreements, οι οποίες θα πρέπει να βασιστούν πάνω σε εμπειρία. Χρειαζόμαστε κάποιο τρίτο μέρος που θα πιστοποιεί τις ε, υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, ε, όπως γίνεται για παράδειγμα με τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Συμπερασματικά λοιπόν έχω να σας πω το εξή. Είναι ένα μεγάλο βήμα μπροστά, αλλά θα είναι τόσο δύσκολο όσο είναι το να έχει κανείς τα υπολογιστικά μηχανήματα εντός της εταιρείας του και να περάσει σε χρήση υπολογιστικών μηχανημάτων που βρίσκονται κάπου αλλού. Ευχαριστώ. Thank you. Thank you very much for this. Σας ευχαριστώ λοιπόν και για αυτές τις διαστάσεις του προβλήματος που είναι πολύ σημαντικές. Τώρα θα περάσουμε στα πρότυπα και το σύννεφο, η συνεισφορά της έτσι η είναι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων. Ίσως να μην γνωρίζετε το έτσι. Μπορεί να μην είστε λοιπόν ιδιαίτερα ενήμεροι για το έτσι. Είναι καρπός της ευρωπαϊκής πολιτικής το 1988 υπήρξαν τα πρώτα επίπεδα, πρότυπα για τις τηλεπικοινωνίες στα πλαίσια του CEPT. Και όταν χρειάστηκε η Ευρώπη δεύτερης γενεάς πρότυπα, που ισχύουν ακόμα αλλά και έχουν εξελιχθεί βέβαια στα πλαίσια του GSM, δημιουργήθηκε το CEPT, η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών. Είμαστε εν μέρη λοιπόν τα δικά σας παιδιά. Έπρεπε να σας το θυμίσω. Έχω αφήσει και την ετήσια έκθεση της έτσι στην είσοδο αν σας ενδιαφέρει έχει μεγαλώσει πάρα πολύ η έτσι, έχει πολύ πιο ε, μεγάλο ίχνος από ό,τι στο παρελθόν και στις τηλεπικοινωνίες, σταθερές τηλεπικοινωνίες, ραδιοεπικοινωνίες. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι να δει κανείς ότι έχουμε μέλη σε 62 χώρες και για τον έφος βλέπουμε ότι το 80% προέρχονται από την βιομηχανία, από ρυθμιστικές αρχές που συμμετέχουν στον καθορισμό των προτύπων. Και θα ήθελα να πω ότι τα πρότυπα είναι μια υδροπονική εκτός εδάφους θα έλεγα προσπάθεια καθορισμού. Εμείς λοιπόν στην έτσι προσπαθούμε να στηρίξουμε αυτό το πράγμα που βρίσκεται από τη φύση του λίγο στον αέρα. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντόπισε τρεις τομείς ή και τρία εμπόδια αν θέλετε για την διεύρυνση της χρήσης του νέφους. Υπάρχουν τα προβλήματα τα συμβατικά, το νομικό πλαίσιο και υπάρχουν επίσης και αυτό που ονομάζουμε μια ζούγκλα από πρότυπα. Ελέγξαμε λοιπόν σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής και μπορεί ο συνάδελφος της Επιτροπής να με ελέγξει και μας ζήτησε η Επιτροπή να έρθουμε σε επαφή με τους εμπλεκομένους και να εντοπίσουμε μέχρι το 2013 να σχεδιάσουμε ένα λεπτομερή χάρτη των απαραίτητων προτύπων για θέματα διαλειτουργικότητας, ασφάλειας, δυνατότητας μεταφοράς δεδομένων και αντίστροφης μεταφοράς. Το θέμα έτσι όπως το έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έλεγα υπογραμμίζει και τα προβλήματα στα οποία πρέπει να σταθώ. Ο συντονισμός για τον καθορισμό των προτύπων, καταρχάς να πω καλύτερα ότι είμαστε καλοί στα πρότυπα. Ο συντονισμός των προτύπων είναι κάτι το σχετικά καινούριο και για τον έφος και για κάποιους άλλους τομείς. Εμείς μαθαίνουμε προχωρώντας Έχουμε όμως και κάποια ερωτηματικά στα οποία δεν έχουμε δώσει απαντήσεις. Ε, η παρουσίαση που σας κάνω εδώ είναι εμπειρική θα έλεγα, βασίζεται στις εμπειρίες που έχουμε συλλέξει. Όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές και κάτι θα που θα ακούσετε συχνά, δεν ξεκινήσαμε από, ε, από ένα λευκό χαρτί Υπάρχουν ε, ε, ήδη κάποια πρότυπα, υπάρχουν κάποιοι κανόνες, περιορισμοί κτλ. Και για να μπούμε εκεί που είμαστε τώρα χρειάστηκε να κάνουμε μία προσπάθεια. Εμείς λάβαμε υπόψη μας το τοπίο ως έχει. Είναι ένα μεγάλο τοπίο, ένα ευρύ τοπίο, πρέπει να μιλήσει κανείς με τους σωστούς ανθρώπους Εμείς δεν είμαστε σε αυτή τη φάση, σε φάση παραγωγής, είμαστε σε φάση συντονισμού στηρίζοντας τους στόχους των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην αρχή μας λέγανε γιατί τώρα τι ανάγκες έχει η Ευρώπη. Η αγορά είναι παγκόσμια, η αγορά είναι σφαιρική. Προφανώς. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορές, υπάρχουν κενά, αναλύουμε τα κενά και προσπαθούμε να τα καλύψουμε. Αυτό που σημαίνει, αν θέλετε αυτό που λέω τώρα, ε, σκεφτείτε λίγο. Κάποτε λέγαμε θα προχωρήσουμε σε καθορισμό προτύπων α, β, γ μέχρι το ω. Τώρα όμως τέθηκε το θέμα της διαλειτουργικότητας και του συνδυασμού όλων αυτών των προτύπων. Μιλάμε για πράγματα που είναι διαφορετικά από, την, από τα κινητά τηλέφωνα. Πρέπει να διασφαλίσουμε τη διαλειτουργικότητα, πρέπει να κάνουμε ε, τεστ, πρέπει να ε, περάσουμε σε διαδικασίες αδειοδότησης και έγκρισης. Ξεκινήσαμε λοιπόν με τα υπάρχοντα υλικά, αξιολογήσαμε στο τέλος της διαδικασίας τα υλικά αυτά Προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε τα αποτελέσματα αυτών των προσπαθειών για να έχουμε ένα πρώτο σταθερό θα έλεγα σημείο. Τώρα σχετικά με τον έφος, μιλάμε για ένα γλυκό με πολλές στρώσεις. Υπάρχουν απαιτήσει, υπάρχουν προβλέψεις, υπάρχουν εμπορικές συμβάσεις, υπάρχουν συμφωνίες για την παροχή ενός κάποιου επίπεδου υπηρεσιών κτλ. Να σας εξηγήσω λίγο ανεκδοτολογικά. Στην πρώτη συνάντηση του έτσι για το συγκεκριμένο θέμα, και αυτό δεν είναι εμπορικό μυστικό, όχι μάλλον και είναι. Είχαμε τον ε, διευθύνοντα σύμβουλο μιας μεγάλης ε, γερμανικής αεροπορικής εταιρείας της οποίας το όνομα ξεκινάει με «ΕΛΑ» και μας είπε ότι τα δεδομένα των πελατών μας είναι το μεγαλύτερο αν θέλετε σημείο του ενεργητικού μας και απαιτείται να υπάρχει μια απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων πριν περάσουμε στον έφος και δεν θα περάσουμε στον έφος αν δεν είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Οι ε, παροχή υπηρεσιών μας είπαν μη σας νοιάζει, οι μηχανικοί μας δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο και θα σας δώσουν τις λύσεις που ε, ε, που χρειάζεται. Κοιτάξτε, είπαμε, εγώ είμαι ο πελάτης. Αν δεν κάνετε αυτό το οποίο θέλουμε να κάνετε, δεν χρησιμοποιούμε τον έφος. Μιλάμε λοιπόν για δημιουργικότητα, μιλάμε για την εμπορική διάσταση, μιλάμε για την ανταλλαγή υπηρεσιών και συνδυασμός διαφορετικών επιπέδων, συνδυασμός αν θέλετε των διαφορετικών στρωμάτων που συναποτελούν αυτή την κατασκευή. Εξορισμού λοιπόν ε, καμία οργάνωση καθορισμού προτύπων δεν μπορεί να το κάνει η μόνη της. Κανένας δεν έχει την αρμοδιότητα να αποφασίσει για τη συνδεσιμότητα, για τις εμπορικές συμβάσεις, για την τεχνική υποστήριξη, για τη συντήρηση των δικτύων. Γενικά όλα αυτά απαιτούν συντονισμό. Ήταν και αρκετά ενδιαφέρον το θέμα αυτό όταν το αντιμετωπίσαμε για πρώτη φορά. Το τρίτο θέμα ίσως είναι και το πιο σημαντικό. Αν πράγματι υπάρξει ένας χάρτης αυτών των standards, αυτών των προτύπων και κάνει κανείς μια ανάλυση αυτών των προτύπων και αυτό το κάνουμε σε απόκριση αν θέλετε των ετοιμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το θέμα δεν είναι τα πρότυπα, δεν είναι ε, οι ε, τεχνικές ρυθμίσεις, αλλά η ικανοποίηση των απαιτήσεων των χρηστών. Αυτό ήταν το θέμα, όπως επίσης και το επιχειρηματικό αν θέλετε κομμάτι. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί κανείς να δει τι τεχνολογίες θα χρειαστεί και τι συνδυασμό τεχνολογιών θα πρέπει να προχωρήσει. Οι απαιτήσει των πελατών λοιπόν είναι πρώτες και η τεχνολογία και τα πρότυπα ακολουθούν. Αυτό που σημαίνει η προσπάθεια που κάνουμε είναι η εξή: είναι η συνεργασία ισότιμη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ε, εξεπλάγημεν στην αρχή όταν είδαμε από πλευράς των κρατών μελών διάφορες αντιδράσεις. Όχι γιατί αυτό θα κόστιζε κάποια χρήματα επιπλέον, αλλά γιατί έβλεπαν ότι υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις στον τομέα του νέφους και είχαν δισταγμούς να τη συζητήσουν με το ιδιωτικό τομέα, με τους εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα. Τίθεται εδώ μια ενδιαφέρουσα ερώτηση και τη θέτω. Ως έχει, αν έχετε την απάντηση να μου την πείτε. Ας πούμε, ιδιωτικότητα, προστασία προσωπικών δεδομένων, τι πολιτική θα ακολουθήσουμε. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μέχρι τώρα οι ρυθμίσεις ισχύουν σε περιφερειακό επίπεδο. Δεν είναι ίδιες στην Κίνα, δεν είναι ίδιες με αυτές της Ευρώπης. Γνωρίζουμε ότι η βιομηχανία, ο τομέας αυτός δεν θέλει να υπάρχουν διπλά επίπεδα και διπλές απαιτήσει και πρότυπα. Πόσο σφαιρικά πρότυπα θα μπορούμε εμείς να παράγουμε όταν οι απαιτήσει των πελατών χαρακτηρίζονται από το περιφερειακό τους χαρακτήρα. Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση και πρέπει να απαντηθεί. Λοιπόν, τι κάνουμε. Ξεκινήσαμε κάτι το οποίο ε, ονομάζεται ε, Cloud Standards Coordination. Ξεκινήσαμε πέρυσι η προϋπόθεση της Επιτροπής είπε να ήταν ανοιχτή αυτή η διαδικασία, πράγματι ήταν ανοιχτή, συμμετείχαν πάρα πολλές οργανώσεις χρηστών, επαγγελματικές, εργοδοτικές και οι δικοί σας, ερευνητικά κέντρα. Γίναμε παγκόσμιοι ε, ξεκινώντας από το μηθέν, συνεργαστήκαμε και με τους Ιάπωνες ρυθμιστές αντίστοιχων πολιτικών, δημιουργήσαμε μία στρόφιγγα επικοινωνίας και αλληλοτροφοδότησης με την πλατφόρμα ε, που συγκεντρώνει όλους όσους ενδιαφέρονται και εμπλέκονται στα θέματα της πληροφορικής και της ε, ε, τηλεπικοινωνίας. Είναι το λεγόμενο ICT Multi-Stakeholder Platform. Είπαμε ότι θα δώσουμε τα σχέδια αυτά στο τέλος του επόμενου μήνα και στο τέλος του χρόνου θα έχουμε τα τελικά αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής. Και τα μέλη του έτσι έχουν συνεισφέρει ιδιαίτερα. Αυτό ήταν το πρόγραμμα. Σε επίπεδο εκτέλεσης του προγράμματος δημιουργήσαμε μια δικτυακή πλατφόρμα, δημιουργήσαμε ένα ηλεκτρονικό χώρο εργασίας, Ε, με τέτοια ένταση στην εργασία μας ο ηλεκτρονικός τόπος συνεργασίας ήταν ο καλύτερος. δημιουργήσαμε συγγνώμη, τρία επίπεδα, τρία ομάδες εργασίας, συν μία ομάδα αναφοράς, σχεδόν 300 είναι αυτοί που συμμετέχουν στην προσπάθεια. Ε, τα αποτελέσματα της ομάδας εργασίας 1 και 2 είναι έτοιμες και περιμένουν να συνδεθούν και με τα αποτελέσματα της ομάδας εργασίας 3 έτσι ώστε να έχουμε την πρώτη απάντηση στο τέλος του μήνα. Προχωράμε έγκαιρα, προχωράμε σωστά και τα αποτελέσματα αν θέλετε έχουν ήδη, είναι ήδη μπροστά μας. Ε, τελικά όλα αυτά θα φανούν αναλυτικά όταν δώσουμε αυτούς τους χάρτες της χρήσης ε, των προτύπων των νεφών, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μιλάμε για διαστημική επιστήμη εδώ, είναι συγκεκριμένα τα πράγματα που έχουμε στη διάθεσή μας. Το πολιτικό μήνυμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν ένας κρίσιμος παράγοντας, μας έδειξε ποιοι είναι οι παράγοντες τους οποίους θα εντάξουμε σε αυτή την ιστορία. Λόγω ακριβώς ε, της συμμετοχής των οργανώσεων των προσώπων των περιφερειών που συμμετέχουν είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει όχι μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ευρωπαϊκά σε εισαγωγικά νέφη, αλλά είναι κάτι το οποίο θα είναι χρήσιμο σε παγκόσμιο επίπεδο για τα πρότυπα λειτουργίας των εφών. Και τέλος, αν δείτε ότι υπάρχουν και άλλοι τομείς των οποίων οι κώδικες προτύπων συμπίπτουν, εδώ θα παίξουμε ένα κάποιο ρόλο. Μερικές φορές σε ορισμένους τομείς υπάρχει τεχνολογία, σε άλλους τομείς όχι. Συνεργαζόμαστε με αυτούς τους τομείς Αυτό το πρότυπο το οποίο εμείς θα καταλήξουμε είναι κάτι το οποίο θα παίξει ένα θετικό ειδικό ρόλο σύγκλησης. Λοιπόν, για μια ακόμη φορά ε, θα μοιραστούμε μαζί σας την προσπάθεια την πειραματική που κάνουμε. Έχουμε ήδη τα πρώτα προϊόντα, τους πρώτους καρπούς. Δύσκολο το βήμα, απαραίτητο όμως. Και για πολλούς άλλους τομείς και όχι μόνο για τα νέφη. Σας ευχαριστώ και τώρα για θέματα ασφάλειας ε, του νεφους έχουμε τον ε, δόκτωρα Γιώρης Φον Χομπουκέν από το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση. Είμαι ο Γιώρης Φων Χόμποκεν, ναι, είμαι νομικός σύμβουλος στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ και είμαι ειδικό σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη ρύθμιση σε ό,τι αφορά την ελευθερία της έκφρασης στο διαδίκτυο, την ασφάλεια του διαδικτύου και το καθεξής. Ε, θα σας μιλήσω για μια έρευνα που έγινε στο ε, Ίδρυμα Έρευνας για ένα θέμα που άπτεται της ασφάλειας ε, των προσωπικών δεδομένων και της προσωπικής σφαίρας των δεδομένων σε ό,τι αφορά τη μετάβαση στον έφος. Δεν είμαι τεχνικός, αν και έχω κάποιο τεχνικό υπόβαθρο, ούτε πρόκειται να μιλήσω για τεχνικά ζητήματα, ξέρετε. Είμαι νομικός ε, και κυρίως πολιτικά ζητήματα και νομικά ζητήματα θέλω να θίξω. Είναι σαφές, θεωρώ, βλέποντας αυτή τη μετάβαση και σε οργανωτικό και σε προσωπικό επίπεδο, όλοι ανησυχούμε για το τι συμβαίνει στα προσωπικά μας δεδομένα όταν αποθηκεύονται στον έφος. Και γι' αυτό θα σας μιλήσω στην παρουσίασή μου. Αυτό θέτει πολλά και ευαίσθητα ζητήματα. Κάποια εξ αυτών να τα ανέφεραν και οι προηγούμενοι ομιλητέ. Πώ θα οργανωθεί η ασφάλεια, για παράδειγμα, στο περιβάλλον αυτό. Εγώ θα μιλήσω για ένα από αυτά τα θέματα για το οποίο ως ακαδημαϊκοί και ερευνητέ θεωρούμε ότι χρειάζεται πιο πολύ έλεγχο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το θέμα της ευαλωτότητας ε, των δεδομένων και η πρόσβαση από τις αλλοδαπές κυβερνήσεις. Και αυτό μας φέρνει στο Patriot Act, αυτή τη συζήτηση για το επίμαχο αυτό ζήτημα, το αμερικανικό αυτόν νόμο. Θα σας εξηγήσω περισσότερα γι' αυτό. Είμαι ακαδημαϊκός ερευνητής. Μας ζητήθηκε λοιπόν να εξετάσουμε κατά πόσον στέκουν οι ανησυχίες του κοινού για το Patriot Act και σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα τη μετάβαση ε, της επιστημονικής έρευνας στον ε, Ολλανδικού κλάδο στον ΕΦΟΣ το εξετάσαμε γιατί σε επίπεδο πανεπιστημίων υπάρχει η ανησυχία ότι αν περάσουμε στον έφος και αν χρησιμοποιήσουμε κάποιες υπηρεσίες τέτοιων ε, παρόχων, ε, εκτιθέμεθα σε τέτοια προβλήματα. Αυτό προβάλλεται και στα μέσα ενημέρωσης και ακόμα και άνθρωποι που δεν είναι ειδικοί ανησυχούν και φυσικά οι πολιτικοί ηθήνοντες ανησυχούν. Όπως για παράδειγμα βλέπουμε ότι και ο CEO της Lufthansa έχει τέτοιες ανησυχίες. Το εξετάσαμε λοιπόν το θέμα αυτό και καταλήξαμε σε τέσσερις ε, πελάτες ε, υπηρεσιών νέφους και ότι όντως αυτή η μετάβαση στις υπηρεσίες νέφους ε, οδηγεί σε μείωση όντως του επίπεδου ασφάλειας ή του ελέγχου του επίπεδου ασφάλειας. Και ιδιαίτερα σε αυτό το πρόβλημα πρόσβαση σε, σε δεδομένα από αλλοδαπές κυβερνήσεις. Αυτό ήταν το βασικό πόρισμα της έρευνας και καλύφθηκε εκτενώς ε, στον διεθνή τύπο. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρουσιάσω ποιο είναι το πρόβλημα. Ένα πρώτο παράδειγμα. Η ηλεκτρονικά δεδομένα και αποθήκευσή τους. Πρόκειται για ένα ζήτημα, ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο πέρασε το 2006 το Κοινοβούλιο. Μετά από πολλή συζήτηση για το κατά πόσο ήταν καλή ιδέα ή όχι, η συζήτηση αυτή εκτελήσεται ακόμα, δεν πρόκειται να επισέλθω σε λεπτομέρειε, αλλά ουσιαστικά τι σημαίνει ότι τα δεδομένα τηλεπικοινωνιών, τα δεδομένα τα τοπικά ε, των ε, Ευρωπαίων πολιτών αποθηκεύονται για μήνες, κάποιες φορές ε, και για έτη ολόκληρα. Σε τι συμπέρασμα μας οδηγεί αυτό. Μπορούμε καταρχάς να έχουμε ε, αμφιβολίες για το κατά πόσον είναι σωστό να αποθηκεύονται ή όχι αυτά τα δεδομένα σε πρώτη φάση. Αλλά να δούμε τι θα γίνει αν τα δεδομένα αυτά μεταφερθούν στον έφος. Ενδεχομένω να διαφωνεί κανένα για το κατά πόσο είναι καλή ιδέα η αποθήκευση των δεδομένων αυτών, αλλά όλοι θεωρώ ότι συμφωνούμε ότι τα δεδομένα αυτά δεν θα πρέπει να καταστούν διαθέσιμα σε αλλοδαπέ κυβερνήσει. Αυτό μου φαίνεται λογική απόρρια. Υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Η μετάθεση των δεδομένων αυτών στον έφος θα μπορούσε να σημαίνει πρόσβαση σε αυτά από ε, πες κυβερνήσεις ε, χωρίς τις απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες. Δυστυχώς, το πόρισμα της έρευνα είναι ότι ναι, κάτι τέτοιο ισχύει. Ιδιαιτέρως, τι εξετάσαμε, ένα νόμο που ισχύει στις ΕΕΠΑ που πέρασε το 2008 που δίνει ε, τέτοια δυνατότητα πρόσβασης σε δεδομένα άλλων δαπών πολιτών. Είναι το FISA Amendment Act. Άρα η απάντηση στην ανησυχία αυτή, ναι, είναι καταφατική. Μας ανησυχεί πραγματικά αυτό. Ένα άλλο παράδειγμα. Σε αυτή την περίπτωση ηλεκτρονικών δεδομένων ανησυχούμε γιατί ένας πάροχος έχει πρόσβαση σε δεδομένα άλλων πολιτών. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, τα συμφέροντα ε, μιας οργάνωσης. Ας εξετάσουμε μια υποθετική περίπτωση, δεν ξέρω καν από το πώς ισχύει, ένα Ολλανδικό Υπουργείο, το Υπουργείο Εξωτερικών, ε, ότι που θέλει να μεταφέρει τα δεδομένα του στον έφος. Όπως καταλαβαίνετε υπάρχει και θέμα απόρριτου διπλωματικών στοιχείων, στοιχείων που έχουν να κάνουν με τις εξωτερικές υποθέσεις της κυβέρνησης. Ε, έχει λόγο να ανησυχεί η κυβέρνηση της Ολλανδίας σε περίπτωση που διαλέξει να μεταφέρει τα δεδομένα αυτά στον έφος. Θεωρείτε, το πω αλλιώς, θεωρείτε ότι θα ανησυχήσει η Ολλανδική κυβέρνηση και θα ψάξει να βρει ποιον πάροχο θα επιλέξει. Κατά πάσα πιθανότητα ναι. Άρα αυτό μας καταδεικνύει τι κίνδυνος ε, ενέχεται. Τίθεται θέμα λοιπόν αλλοδαπής ε, δικαιοδοσίας. Αυτό δεν είναι θέμα, ξέρετε, σε ό,τι αφορά την τεχνική ε, άποψη. Δεν ε, μιλάμε για κάτι παράνομο, μιλάμε για κάτι νόμιμο σύμφωνα με τους νόμους μιας ξένης χώρας σε ό,τι αφορά την πρόσβαση δηλαδή στα δεδομένα αυτά. Αλλά περιλαμβάνει την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών. Άρα αυτή η πρόσβαση επιτρέπεται ρητά από μια δημοκρατική διαδικασία άλλης χώρας αυτό που έχουμε εξετάσει πιο πολύ είναι το νομοθεσία των ΙΠΑ. Δύο ερωτήσεις λοιπόν θα ήθελα να κοιτάξω ε, περαιτέρω. Ε, ερωτήσεις που δύο συνάδελφοί μου, ο κύριος Άξελ Άντμα και ο κύριος Νίκο Φωνέικ, ε, θα ε, απαντήσουν στη σχετική τους μελέτη, η οποία θα δημοσιευθεί πρόσφατα. Καταρχάς λοιπόν, κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης των δεδομένων αυτών από άλλες ε, κυβερνήσεις. Ε, για παράδειγμα, η κυβέρνηση της ΕΠΑ ζητά πρόσβαση σε δεδομένα ε, πολιτών, Ευρωπαίων πολιτών. Συμβαίνει κάτι τέτοιο όμως. Υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει δυνατότητα μεν, αλλά πρέπει να μας ανησυχεί κάτι τέτοιο. Μια γενική ανάλυση των γενικών τάσεων βάσει της σχετικής ακαδημαϊκής ε, βιβλιογραφίας και των, γενικών, ε, των γενικότερων ε, ερευνών. Διαπιστώνουμε ότι κάτι τέτοιο λοιπόν συμβαίνει. Υπάρχει μια γενική τάση πρόσβασης δεδομένων μέσω των παρόχων του νέφους. και κάποιες κυβερνητικές υπηρεσίες μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματικές σε ό,τι αφορά την ε, υποκλοπή στοιχείων, γιατί ε, σε πολλές περιπτώσεις ε, αποθηκεύονται στον έφος, χωρίς κωδικοποίηση. Αυτό αποτελεί και ένα κίνδυνο. Γιατί αν ισχύει κάτι τέτοιο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστούμε μια τέτοια ε, κατάσταση. Ο αντίκτυπος είναι εντελώς ασαφής. Αυτό που προσπαθούμε είναι να κάνουμε μια ανάλυση για το πώς μπορούμε να το πετύχουμε κάτι τέτοιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για μια οργάνωση να διαχειριστεί ένα τέτοιο κίνδυνο. Και αυτό ασφαλώς αποτελεί πηγή ανησυχία. Αν ε, ξέρει κανείς ότι υπάρχει ο κίνδυνος ε, μεν, αλλά μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με τον χύψη τρόπο, το πρόβλημα είναι πιο περιορισμένο. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα μεγάλο πρόβλημα. Επιπλέον βλέπουμε ότι υπάρχουν και πιο συγκεκριμένες εξουσίες που υπησέρχονται, για παράδειγμα, η αστυνομία, η εθνική ασφάλεια και η οργάνωση όλων αυτών θα πρέπει να συνάδει με την ψηφιακή αυτή μετάβαση. Θα πρέπει να εξυγχρονιστούν οι εξουσίες των σωμάτων αυτών. Και βλέπουμε στη ΣΥΠΑ, έχουμε αυτή το Visa Amendments Act, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες δυνατότητες που επιτρέπουν την πρόσβαση σε τέτοιες υπηρεσίες εξ αποστάσεων, υπολογιστικές υπηρεσίες εξ αποστάσεων, όπως αναφέρονται και στην, στην Ευρώπη θα δούμε ότι θα περάσουν και θα επιβληθούν τέτοιες συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε σε επίπεδο ρυθμιστικό, σε επίπεδο πολιτικής. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θελήσαμε να εξετάσουμε στην έρευνά μας. Μπορούμε φυσικά να το ε, να δώσουμε μια απάντηση μέσω τεχνικών μέσων, με περίπλοκο τρόπο, να προσπαθήσουμε να πετύχουμε ε, δικλείδες ασφαλείας, ε, εγγυήσεις ε, σε ό,τι αφορά τα εθνικά σύνορα κάθε χώρας, αλλά εμείς τι είπαμε, είπαμε ότι ας το εξετάσουμε σαν ένα νομικό πρόβλημα, το οποίο ενδεχομένως να μπορέσει να λυθεί με νομικά μέσα, με κάποιες, με νομοθεσία. Τέσσερις λοιπόν προσεγγίσεις εξετάσαμε. Καταρχάς, κατά πόσον το θέμα αυτό θα μπορούσε να ληφθεί στην δικαιοδοσία όπου προκαλείται το πρόβλημα, δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση στη ΣΥΠΑ. Αυτό συζήτησαμε ιδιαίτερω. Να προσπαθήσουμε να ζητήσουμε να ταποποιηθεί το FISA Amendments Act για να προσθεθούν δικλείτες ασφαλείας που θα εγγυούνται το απόρριτο των προσωπικών δεδομένων των ατόμων που ζουν εκτός ΙΠΑ. Το εξετάσαμε λοιπόν αυτό ως ενδεχόμενο και κοιτώντας κατά πόσον είναι εφικτό, πολιτικά κυρίως εφικτό κάτι τέτοιο, καταλήξαμε ότι μάλλον δεν υπάρχει εφικτότητα, μάλλον δεν είναι εφικτό κάτι τέτοιο ως ενδεχόμενο. Επίσης εξετάσαμε πρόσφατα τώρα το δικαστήριο των ΗΠΑ, εξέτασε κατά πόσον είναι συνταγματικός καν αυτός ο νόμος, το Visa Amendment Act και αποφάνθηκε το δικαστήριο ότι ούτε καν οι Αμερικανοί δεν είχαν δικαίωμα να ασκήσουν, να καταγγείλουν τέτοια ζητήματα για τον νόμο αυτό. Ένα δεύτερο θέμα, το οποίο ανέφερε και η Επιτροπή Ρέντινγκ, έχει να κάνει με το διεθνές δίκαιο. Νομίζω ότι υπάρχει αυτή η ιδέα ότι υπάρχει κυριαρχία ε, των, επί των δεδομένων κάθε χώρας υπάρχει, ας θέλετε, αυτή η αίσθηση της ε, διαμεθοριακής κατασκοπίας. Αν κοιτάξουμε λοιπόν το θέμα αυτό σε επίπεδο εθνικής ασφάλειας, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στα δεδομένα στο εξωτερικό, στην Αλλαδαπή, σε άλλη δικαιοδοσία, διαπιστώνουμε ότι δύσκολα μπορούμε να χειριστούμε κάτι τέτοιο. Υπάρχουν μεγάλες αμφιβολίες κατά πόσον το διεθνές δίκαιο θα δικαιολογούσε μια τέτοια καταγγελία ενδεχομένως στο Διεθνές Δικαστήριο. Δεν είμαι απόλυτα ειδικό σε τέτοια θέματα, αλλά δεν θεωρούμε ότι θα ήταν επιτυχής μια τέτοια καταγγελία. Κάτι άλλο τώρα. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα το αναφέρω στα καταληκτικά μου σχόλια. Αλλά εξετάσαμε κατά πόσον αυτό θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο κράτους μέλους. Και τελικά καταλήγουμε στο ότι ναι, αυτό θα είχε νόημα. Ιδιαίτερο, εξετάζοντας τι μας λένε οι εθνικές μυστικές υπηρεσίες, τι κάνουν οι εθνικές μυστικές υπηρεσίες σε κάθε χώρα που ενδεχομένως ανησυχεί για κάτι τέτοιο. Στις κατοχώρες βλέπουμε ότι στην ετήσια έκθεση των μυστικών υπηρεσιών εκφράζεται μια συγκεκριμένη ανησυχία σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Πρόκειται φυσικά για ένα παράγοντα έκθεσης της χώρας. Και όχι μόνο της δικής μας χώρας, αλλά και άλλων χώρων. Και έτσι βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη συμφωνία σε επίπεδο Ολλανδικών Μυστικών Υπηρεσιών. Θεωρείται ότι υπάρχει πρόβλημα, πραγματικά. Ίσως, λοιπόν, επί της βάσης αυτής κάτι πιο ενδιαφέρον θα μπορούσε να γίνει. Κλείνοντας, να πω δύο λόγια για το ευρωπαϊκό επίπεδο, για το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δύο ε, είναι, αν θέλετε, τα σημεία στα οποία διεξάγεται σχετική συζήτηση καταρχάς, ε, ο κανονισμός για την προστασία των δεδομένων και κατά δεύτερον η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απελευθέρωση του πλήρους δυναμικού του νεφούς. Κοιτώντας λοιπόν ε, πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα μέσω της ε, οδηγίας για την προστασία των δεδομένων, Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Το πιο βασικό πρόβλημα όμως είναι ότι το θέμα μας δεν είναι μόνο θέμα προσωπικών δεδομένων. Είναι θέμα διαχείρισης απορρίτου και έχει να κάνει και με την ε, οργανωτική ασφάλεια, τα στρατηγικά συμφέροντα κυβερνήσεων, επιχειρήσεων. Όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν με την διαχείριση προσωπικών δεδομένων και επιπλέον θα πρέπει να αναρωτηθούμε Ποια είναι η αξία του πλαισίου ε, προστασίας δεδομένων σε ό,τι αφορά την ε, διασφάλιση του απορρίτου και της εμπιστευτικής σφαίρας. Δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειε, αλλά πιστεύω ότι δεν είναι αυτό το σωστό πλαίσιο για να διασφαλίσουμε το απόρριτο των δεδομένων. Έχει να κάνει με την ροή των προσωπικών δεδομένων, όχι με το απόρριτο των προσωπικών δεδομένων. Άρα, δεν μας καλύπτει το πλαίσιο αυτό. Όχι υπαρκώς, σε πάση περιπτώσει. Κοιτώντας τι γίνεται στο πλαίσιο αυτό, με την ανακοίνωση για την απελευθέρωση του δυναμικού του νεφούς. Υπάρχουν εδώ κάποιες αναφορές στο θέμα αυτό, αλλά περιορίζονται σε ό,τι αφορά θέματα εφαρμογής του νόμου. Δεν αναφέρονται αρκετά όλες οι πτυχές του προβλήματος και πώς θα πρέπει να τις διαχειριστούμε. Αυτό μας ανησυχεί. Νομίζω ότι στο σημείο αυτό θα πρέπει να ολοκληρώσω. Θα δεχτώ ερωτήσεις. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκτός μικροφώνου η κυρία Πρόεδρο, η κυρία Ομιλήτρια. Good afternoon and... Καλησπέρα σας. Ε, ευχαριστώ πολύ που καλέσατε και την πλευρά των καταναλωτών ε, σε αυτή την ακρόαση. Εγώ εκπροσωπώ την ΜΠΕΚ, την Οργάνωση Ευρωπαϊκών Καταναλωτών και αντιπροσωπεύουμε 41 εθνικές οργανώσεις καταναλωτών. Και θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι από τις αρχές συμφωνούμε απόλυτα ότι οι εξελίξεις στην τεχνολογία απολογιστικού νέφους μπορούν και ήδη μάλιστα παρέχουν πολλά πολύ αριθμό ωφέλη στους καταναλωτές. Όπως είπαμε προηγουμένως, οι καταναλωτές όλο και περισσότερο χρησιμοποιούν το υπολογιστικό νέφος για τα δεδομένα τους και τις υπολογιστικές τους εργασίες, ξεκινώντα από τις δικέ τους συσκευές. Τα ωφέλη αναφέρθηκαν ήδη από τον προηγούμενο μιλητή από την Τελεφώνικα, και αφορούν τη μεγαλύτερη χωρητικότητα αποθήκευσης, μεγαλύτερη ευκολία, εύκολη πρόσβαση σε πολλές υπηρεσίες και σε δεδομένα και επίσης το υπολογιστικό νέφος θα προσφέρει μάλλον ελπίζουμε μεγαλύτερη αξιοπιστία και προστασία των δεδομένων των καταναλωτών και θα μπορούσε επίσης να παράσχει ενδιαφέροντες καινοτόμους τρόπους αλληλεπίδρασης με τους άλλους ανθρώπους. Από την άλλη όμως γνωρίζουμε ότι παρουσιάζει και σημαντικούς κινδύνους για τους καταναλωτές όταν αυτοί βάζουν την προσωπική του ζωή στο υπολογιστικό νέφος. Αναφέρθηκαν ήδη ορισμένοι κυριακοί κίνδυνοι. Ε, τίθενται κάποιοι κίνδυνοι προσωπικών δεδομένων, έλλειψη ελέγχου των προσωπικών δεδομένων καθώς και ανεπαρκείς πληροφορίες για τους καταναλωτές όσον αφορά το πώς, πού και από ποιον φυλάσσονται τα δεδομένα ποιος είναι ο ιδιοκτήτης τους. Και ο δεύτερος κίνδυνος που θέλω να επισημάνω σήμερα και που αναφέρεται στη στρατηγική είναι η πιθανή χρήση αθέμητων άδικων όρων συμβάσεων που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τους καταναλωτές λόγω απώλειας δεδομένων ή άλλων ανεκτημάτων. Πώς απαντάμε εμείς στη στρατηγική της Κομισιόν η ίδια η στρατηγική προφανώς ε, είναι ευπρόσδεκτη ως πρωτοβουλία και απαραίτητη, αλλά κατά την άποψή μας δεν είναι έπαρκος φιλόδοξη. Δεν αντιμετωπίζει ικανοποιητικά αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό για τους καταναλωτές. Και πρέπει να πούμε ότι η πίστη των καταναλωτών είναι αναγκαία για να δεσμευτούν στο περιβάλλον του υπολογιστικού νέφους και αν δεν είναι βέβαιοι ότι θα αποτελέσει για αυτούς θετική εμπειρία, δεν πρόκειται να το πράξουν. Συνεπώς και πάλι αυτό που θεωρούμε εμεί ότι λείπει από τη στρατηγική είναι η καθοδήγηση για τα πιο σημαντικά ζητήματα καταναλωτών που έχουν σημασία στο υπολογιστικό νέφος. Θα σα εξηγήσω αυτό τώρα πιο λεπτομερό Το πρώτο ζήτημα. Είναι ότι έχουμε μια πολύ βαθιά ανησυχία όσον αφορά την δράση κλειδί αριθμό 2 της στρατηγικής σε σχέση με την προστασία από τους ε, ε, ανεπαρκείς κανόνες ε, συμβάσεων και επίσης και τα μέτρα για την προστασία από παράνομες δραστηριότητες ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι οι καταναλωτές θα μπορέσουν να υποφεληθούν στο μέγιστο βαθμό από την ενιαία ψηφιακή αγορά έρχομαι στο πρώτο μου σημείο τους ασφαλείς και δίκαιους όρους συμβάσεων για τους καταναλωτές. Ξέρετε ότι υπό τη δράση κλειδί 2 η Κομισιόν προτείνει μέτρα ώστε να βεβαιωθεί ότι θα διασφαλίζονται ασφαλείς και δίκαιες συμβάσεις για τις υπηρεσίες υπολογιστικού νεφού. Η ανάλυση της Κομισιόν αληθεύει κατά την άποψή μας. Περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση ως χαρακτηριζόμενη από έλλειψη νομικής βεβαιότητας, πολλούς ε, όχι σωστούς όρους συμβάσεων και εκτενής ε, ε, αποποίησης ευθυνών. Αυτοί λοιπόν οι όροι που επιβάλλονται στους καταναλωτές οδηγούν σε απολέμπεις του είναι στις ψηφιακές υπηρεσίες και σε επιφυλάξεις χρήση αυτών των υπηρεσιών. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα. Αλλά τι προτείνει η Κομισιόν για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα πρώτα απ' όλα αναφέρονται στον προτείνομενο κανονισμό για ένα κοινό ευρωπαϊκό νόμο των πολίσεων που ακόμη εκκρεμεί και είναι κρίμα που η κυρία Μπέριγκερ από την Επιτροπή Γιούρη δεν βρίσκεται εδώ επειδή είναι η επί της ουσίας Επιτροπή για το ζήτημα προτείνουν ένα συμπληρωματικό εργαλείο για το δίκαιο των συμβάσεων δηλαδή θα πρέπει να υπάρχουν μοντέλα, υποδείγματα συμβάσεων για τις συναλλαγές αυτές των καταναλωτών που θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους οργανισμούς καταναλωτών και από τη βιομηχανία. Δεν αναφέρονται όλοι αυτοί δυστυχώς μέσα στη στρατηγική. Φαίνεται να είναι καλοσχεδιασμένο σχέδιο, αλλά είναι πολύ ανεπαρκής λύση για τους καταναλωτές. Για ποιο λόγο, διότι ο τρόπος με τον οποίο σκοπεύει να προστατεύσει τους καταναλωτές από αθέμητους όρους η Κομισιόν είναι εθελοντικό. Διότι μιλάμε για αυτόν τον κοινό νόμο πωλήσεων στην Ευρώπη που είναι προαιρετικός. Είναι κάτι, ένα νέο αποκοίημα το οποίο προτείνει η Κομισιόν, ένας νόμος που θα υπάρχει παράλληλα με την υπάρχουσα νομοθεσία σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και αυτό κατά την αποψή μας σημαίνει ότι η Κομισιόν με κάποιο τρόπο ε, μεταθέτει την προστασία των καταναλωτών που είναι απαραίτητη την μεταθέτει και την μετατρέψει σε μια παρά, παράλογη έννοια. Εξαρτάται δηλαδή από τις υπηρεσίες, από τις επιχείρησεις που παρέχουν τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους να αποφασίζουν κατά πώς θα χρησιμοποιούν τους απαραίτητους κανόνες για το υπολογιστικό νέφος. Δηλαδή κατά πώς θα χρησιμοποιούν αυτούς τους προαιτικούς κανόνες ή κατά πώς θα χρησιμοποιούν τους σημερινούς ε, μη εξυγχρονισμένους νόμους που δεν αφορούν συγκεκριμένες ε, περιπτώσεις και που δεν προστατεύουν πραγματικά τους καταναλωτές και είναι Και το θέμα είναι ότι ε, αν οι καταναλωτές ε, δεν καταλαβαίνουν απόλυτα, αυτό σημαίνει ότι δεν λαμβάνουν επαρκή προστασία. Επιπλέον, θα έχουμε κι άλλο ένα προαιρετικό εργαλείο, των Κοινό Ευρωπαϊκό Νόμο για τις ένα πρόσθετο εργαλείο και τις διάφορες συμβάσει. Για να υπάρχει νομική βεβαιότητα που θα θέλαμε όλοι να υπάρχει, νομική ασφάλεια, αυτό πραγματικά είναι ένα δρόμο που θα πρέπει να αποφύγουμε, διότι έτσι θα διαδοθούν πολλά προαιρετικά εργαλεία, συν οι εθνικέ νομοθεσίε και όλα αυτά θα τα έχουν στη διάθεσή του οι επιχείρησει και θα μπορούν να διαλέξουν ό,τι επιθυμούν. Για να κλείσω αυτό το σημείο. Πιστεύω ότι υπάρχει χρόνο ακόμα να αλλάξουμε αυτή την κοινή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των Πολίσεων που εκκρεμίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχουν τροπολογίε που αποσκοπούν στο να μετατραπεί σε οδηγία για τους καταναλωτές. Ε, αυτό πιστεύουμε εμείς ότι θα είναι πολύ πιο χρήσιμο και όχι επιβλαπές, αλλά μάλλον ένα βήμα προς τα εμπρός. Πιο βραχυπρόθεσμα για να μην υπάρχει ο προαιρετικός κανονισμός, εμείς θεωρούμε ότι καλό θα ήταν να υπάρχει κάποια καθοδήγηση για τη χρήση της οδηγίας αθέμητων όρων συμβάσεων που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και πολλά χρόνια, ειδικότερα για τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους. Θα μπορούσε λοιπόν να δώσει κάποια καθοδήγηση η Επιτροπή για τον τρόπο αξιολόγησης ορισμένων ρητορών και να θεσπίσει κανόνες προστασίας ε, ε, με τους οποίους θα μπορούν ε, να ορίζεται κατά πόσο οι κανόνες προστασίας των δεδομένων είναι αθεμητοί ή όχι. κατά πόσο τηρούνται οι απαραίτητοι κανόνε. Το επόμενο σημείο είναι κάτι που αναφέρθηκε ήδη πολλές φορές. Αφορά την προστασία των δεδομένων. Ξέρουμε από τη δική μας εμπειρία ότι η έλλειψη της εμπιστοσύνης των καταναλωτών αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην εξέλιξη της ψηφιακής οικονομίας και η στρατηγική της Κομισιόν επισημαίνει ότι η νομοθεσία προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκκρεμεί αυτή τη στιγμή αποτελεί εργαλείο κλειδί για να υπάρχει εμπιστοσύνη των καταναλωτών για την προστασία των δεδομένων τους και των αναγκών τους από τις επιχειρήσεις. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό και σε αυτή τη συζήτηση να υπογραμμίσουμε ότι η καινοτομία θα μπορέσει να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί σε ευρία κλίμακα μόνο εφόσον οι άνθρωποι έχουν εμπιστοσύνη ότι τα προσωπικά του δεδομένα τη χάνουν τη σωστής διαχείριση. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό αυτή η νομοθεσία, η αναθεώρηση τη νομοθεσία προστασία των δεδομένων να γίνει σωστά. Σε σχέση με τα όσα είπε ο προηγούμενο ομιλητή από την Τελεφώνικα θα ήθελα να αναφέρω ότι χρειάζεται ένα σταθερό, στιβαρό πλαίσιο προστασία δεδομένων στην Ευρώπη για να δημιουργήσει ένα τεράστιο, πιστεύουμε, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει και τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Εν συντομία, θα ήθελα να σα επισημανώ ορισμένα σημεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την αναθεώρηση του νόμου προστασία των δεδομένων. Θα είμαι σύντομη, αλλά παρόλα αυτά σίγουρα η διαφάνεια είναι πάρα πολύ σημαντική για του καταναλωτέ, επειδή πρέπει να γνωρίζουν τι γίνονται τα προσωπικά δεδομένα στο υπολογιστικό νέφο. Το πρόβλημα, όπως το γνωρίζετε και από τη δική σα εμπειρία, είναι ότι με τι προηγούμενε πολιτικέ σε σχέση με τι υπηρεσίε υπολογιστικού νέφους ε, περιλαμβάνονταν πολύ περίπλοκοι όροι τεχνικοί που συχνά δεν συμμορφώνονται με τι αρχέ τη δικαιοσύνη και της διαφάνειας και που δεν ενημερώνουν επαρκώ του καταναλωτέ για το τι συμβαίνει, τι τύχη έχουν τα δεδομένα του. Γράφονται ουσιαστικά για να αποποιούνται οι παροχή της ευθύνες τους ή για την τήρηση ορισμένων απαιτήσεων. Συνεπώς είναι πολύ σημαντικό ο καταναλωτή να καταλαβαίνει κατά πόσο τα δεδομένα του ε, στέλνονται και σε άλλους παρόχους ή σε τρίτα μέρη. Ποια είναι αυτά τα τρίτα μέρη και τι σκοπό έχουν, πώς σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα και ούτω καθεξής. Συνεπώς, οι πολιτικές ιδιωτικού απορρίτου πρέπει να γράφονται με τρόπο τέτοιο ώστε να είναι κατανοητές προς τους καταναλωτές, να περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες, να εξηγούν αυτό που έχει σημασία για τους καταναλωτές. Σας ζητάμε λοιπόν να υποστηρίξετε αυτές τις διατάξεις που έχουμε σε αυτήν την αναθεώρηση της νομοθεσίας προς των δεδομένων που αποσκοπούν ουσιαστικά στο να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια σε σχέση με τις πολιτικές ιδιωτικού απορρίτου. Πολύ σύντομα τώρα η ισχύουσα νομοθεσία οι καταναλωτέ πρέπει να είναι βέβαιοι ότι θα προστατεύονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, από τα ευρωπαϊκά πρότυπα και όχι από οι υπεράκτης δικαιοδοσίες που θα έχουν επιλέξει επιχειρήσεις για να παρακάμπτουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αυτό που χρειαζόμαστε λοιπόν είναι να είμαστε βέβαιοι ότι τα ευρωπαϊκά πρότυπα θα είναι εκείνα που θα εφαρμόζονται στους Ευρωπαίους καταναλωτές στον τομέα του υπολογιστικού νέφους. Το οποίο ακριβώς είναι ανεξάρτητο τοποθεσιών, είναι κάτι δύσκολο συνεπώς, αλλά παραμένει πολύ σημαντικό. Το επόμενο ζήτημα είναι η επιβολή του νόμου στο οποίο αναφέρθηκαν οι προηγούμενοι ομιλητέ, να υπογραμμίσω ότι οι καταναλωτέ σίγουρα φοβούνται και πρέπει να είναι βέβαιοι ότι τα προσωπικά του δεδομένα που μπαίνουν στο υπολογιστικό νέφος δεν θα καταλήξουν σε κάποια ξένη δίκηση, σε κάποια ξένη κυβέρνηση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και τέλο, αυτό που αναφέρει και η Κομισιόν, θα πρέπει να υπάρχει ένα κώδικα διοντολογία για τη βιομηχανία όσον αφορά την εφαρμογή τη προστασία των δεδομένων στο υπολογιστικό νεφο. Θεωρούμε ότι τη θεωρία είναι καλή ιδέα, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν ελάχιστα πρότυπα σε περίπτωση που έχουμε αυτού του κώδικε. Συνεπώ πρέπει να παρακολουθούνται οι επιχειρήσει, να υπάρχουν κυρώσει σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά, να υπάρχει μηχανισμό επίλυση χειρισμού παραπώνων των καταναλωτών και να είμαστε βέβαιοι ότι θα επιβληθεί αυτός ο κώδικας από τις αρχές ε, προστασίας των δεδομένων. Το επόμενο σημείο αφορά τη φορητότητα δεδομένων. Για να έχουμε μια φορά υπολογιστικού νέφους για τους καταναλωτές, η φορητότητα και η κινητικότητα του πελάτη είναι πολύ σημαντική. Αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι σε περίπτωση που αποτύχουν οι στρατηγικές να υλοποιήσουν τα σωστά μέτρα, δεν θα είναι επιτυχής η υπηρεσία. Θέλουμε να αποφύγουμε τον αποκλεισμό, μάλλον τον περιορισμό σε αδιέξοδο των καταναλωτών λόγω κάποιων συμβάσεων, για παράδειγμα, τη δέσμευσή τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα που πρέπει να σεβαστούν σε μια σύμβαση ή για τεχνικούς λόγους. Πιστεύουμε λοιπόν ότι είναι σημαντικό τα τεχνικά εμπόδια μεταξύ παρόχων παρόμοιων υπηρεσιών υπολογιστικού νεύους και φυσικά υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες υπηρεσίες αλλά για παράδειγμα αν έχουμε μια πλατφόρμα μουσικής και θέλουμε να αλλάξουμε πλατφόρμα μουσικής θα πρέπει να, αυτό να γίνεται εύκολα, να μην υπάρχουν δηλαδή τεχνικά εμπόδια. Επίσης είναι σημαντικό σε σχέση με αυτό να υπάρχει δυνατότητα άμεσης μεταβίβασης των δεδομένων μεταξύ ανταγωνιστικών πλατφόρμων ώστε να μην χρειάζεται να κατεβάζει τα πάντα ο καταναλωτής στη δική του συσκευή για να τα στείλει σε έναν άλλο πάροχο στον οποίο θέλει να αλλάξει. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα σε σχέση με το υπολογιστικό νέφος είναι το copyright, τα πνευματικά δικαιώματα και τα σχετικά ζητήματα. Όπως πολύ συχνά ακούμε, αλλά πιστεύω ειδικότερα για τους καταναλωτές είναι πολύ σημαντικό, το κυρίο πλέον έκτημα του υπολογιστικού νέφους είναι φυσικά η προσβασιμότητα στο ψηφιακό περιεχόμενο. Για να αποκτήσει λοιπόν κανείς πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτό θα πρέπει να μπορεί είτε πρόκειται για μουσική, είτε για οπτικό περιεχόμενο, είτε για βιβλία, θα πρέπει από οποιαδήποτε συσκευή να έχει πρόσβαση από την τοποθεσία της επιλογής του, ανεξαρτήτως της εθνικότητας ή του τόπου διαμονής του καταναλωτή. Για να δώσω εδώ μια γενική παρατηρήση, θα πρέπει να είναι σαφές ότι η έννοια του copyright και της διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων βασίζεται στην εδαφικότητα και εξορισμού ορισμός της σημερινής έννοιας, έτσι όπως έχει σήμερα, δεν συνάδει με το cloud computing. Γίνονται κάποιες εργασίες, αλλά εδώ, παρά το γεγονός ότι η Κομισιόν περιγράφει πάρα πολύ καλά στρατηγική το πρόβλημα των καταναλωτών όσον αφορά τα πραγματικά δικαιώματα, δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και τα σχετικά ζητήματα, δεν έχουμε δει κάποια ισχυρή πολιτική βούληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προτείνει μέτρα τα οποία χρειαζόμαστε τόσο επιγόντως για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι θα τηρούνται όλες οι προβλέψεις για την προστασία των διανοητικών δικαιωμάτων. Και η... τα τέλη, όπως είδαμε, είναι κάτι άλλο που δεν έχει αντιμετωπιστεί ιδιαίτερα. Ο κύριος Βιτορίνο προέδρευσε μια πλατφόρμα για να συζητηθεί το άμεσό μέλλον και οι συστάσεις που υιοθετήθηκαν πρόσφατα ουσιαστικά συνιστούν διαρκή ε, εξαφάνιση επιπέδων στο ψηφιακό περιβάλλον και είναι σημαντικό να επιταχύνουμε όσον αφορά αυτέ τι συστάσει. Τώρα, το τελευταίο σημείο που θα αναφέρω, κάτι που δεν αναφέρεται στη στρατηγική τη Κομισιόν, είναι η ανεξαρτησία του δικτύου, η ουδετερότητα. Δεν το αναφέρει η Κομισιόν και δεν ξέρω γιατί. Ουδετερότητα σημαίνει ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο είναι διαθέσιμο στο δίκτυο θα πρέπει να είναι προσπελάσιμο από οποιονδήποτε, ανα πάσα στιγμή, από οποιοδήποτε σημείο του δικτύου, μέσω οποιασδήποτε συσκευή. Εγώ θέλω να υπογραμμίσω εδώ ότι είναι πραγματικά σημαντικό αυτή η αρχή αυτή η ουδετερότητα να θεωρηθεί πρωταρχική αρχή για τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους. Αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε. Δεν θέλουμε να βρούμε σε μια κατάσταση όπου ορισμένοι υπάρχουν δεν θα σας επιτρέπουν να πάτε στις υπηρεσίες ε, υπολογιστικού νέφους που προτιμάτε. Θέλουμε να αποφύγουμε ένα τέτοιο σενάριο και θα θέλω να κλείσω λέγοντας ότι είναι πολύ σημαντικό η Κομισιόν να συνεχίσει να μελετά αυτό το ζήτημα και να δούμε ε, τις επιπτώσεις αυτές στο ευρύ φάσμα των υπηρεσιών υπολογιστικού Σα Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή uh, σας. ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους τους ομιλητές. Νομίζω ότι είχαμε μια έτσι σχετικά συνολική εικόνα των πραγμάτων. Πάρα πολλοί τομείς συμπεριελήφθησαν και από πλευράς των χρηστών και από πλευράς της νομικής ε, κάλυψης και οι θέσεις ε, του Κοινοβουλίου και για το Κοινοβούλιο ειδικά αυτές οι, οι, ιδέες που ακούσαμε ήταν πάρα πολύ χρήσιμες. Έχουν ζητήσει κάποιοι συνάδελφοι το λόγο. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τον, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι παρούσα σε αυτή τη συνάντηση. Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε λίγο ή να μας μεταφέρετε κάποιες σύντομες σκέψεις. Uh, so please, uh, the floor is yours. So I'll, I'll take the floor because... Είμαι ο τμήματάρχης υπεύθυνο, αυτός που αν γίνει κάτι θα τον πυροβολήσουν. Είτε γιατί δεν τα καταφέρνω στη δουλειά μου, είτε γιατί κάνω λάθη στη δουλειά μου. Σημασία έχει το τελικό αποτέλεσμα βέβαια. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι προοπτικές σας, δεν θα χρειαστώ πολύ χρόνο. Θα μπορούσα όμως γιατί πράγματι έγιναν πάρα πολλές συζητήσεις σχετικά με την τήρηση της τάξης και την ένομη τάξη στο συγκεκριμένο θέμα σχετικά με την πιθανότητα πρόσβαση στα δεδομένα μας από τρίτες χώρες. Αυτό είναι ένα θέμα. Είναι ε, σωστό το ότι δεν το εξετάζουμε λεπτομερώς. Έχει γίνει πολύ γνωστό το θέμα αυτό και στα πλαίσια της έκθεσης της Περσινής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά λόγω και των πολιτικών συζητήσεων που προηγήθηκαν. θα πρέπει να δούμε πώς πράγματι έχουν τα πράγματα. Πρέπει να ισορροπήσουμε τους κινδύνους λίγο. Μην πιστέψετε ότι τα τοπικά πληροφορικά δίκτυα, δίκτυα πληροφορικής είναι ασφαλή από hackers ή από τρίτες χώρες, διότι δεν είναι. Υπάρχει μια κάποια σημασία να μεταφέρει κανείς τα δεδομένα σε πολύ ασφαλή συστήματα από τους πιο ενημερωμένους και προχωρημένους τεχνικούς. Ε, πρέπει να εξορροπήσουμε λίγο, να ζυγίσουμε τους κινδύνους και αυτό το ξεχνάμε. Αναφερθήκατε επίσης και στους παράγοντες μετρίασης σαν τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς οργανωτικούς ή τεχνικούς που έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Η μεγαλύτερη κίνδυνη είναι τα ανθρώπινα λάθη, η μη σωστή εφαρμογή των συστημάτων password, συνθηματικών ονομάτων, Γενικά τα οργανωτικά θέματα έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Υπάρχει επίσης το θέμα του πώς προχωρά στη σύναψη των συμβάσεων. και τα αποτελέσματα αυτά δεν θα πάνε υποχρεωτικά σε, στο δημόσιο νέφος αλλά σε επιμέρους λύσεις ιδιωτικών νεφών. σε κέντρα δεδομένων τα οποία χρησιμοποιούν την τεχνολογία των νεφών. Τώρα δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό αυτό είναι ασφαλές. Και είναι πάρα πολύ πιθανό να μην γνωρίζει κανείς το τι ακριβώς και με ποιο τρόπο λειτουργεί το νέφος. Αυτό είναι θέμα συζήτησης ε, ανάμεσα στην Κίνα και στις Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με τα δίκτυα δεδομένων. Πάντως, τα ευαίσθητα δεδομένα στο μέλλον θα σωρεύονται σε ιδιωτικά σύνολα νεφών ίσως σε κοινέ αν θέλετε προσπάθειες νεφών, δηλαδή κάποιες δημόσιες υπηρεσίες που θα καθορίζουν τα επίπεδα ασφαλείας και όσοι παίρνουν τέτοιες αποφάσεις Έχουμε και συναδέλφους ε, σαν τον συνάδελφο από το Κοινοβούλιο που είναι πάρα πολύ προσεκτικοί γιατί δεν θέλουν να χάσουν τη δουλειά τους. Και εδώ ακριβώς ο κίνδυνος για αυτούς είναι μεγάλος. Πρέπει λοιπόν να πάμε πολύ σιγά, πολύ αργά για να γίνουν τα πράγματα όσο πιο σωστά μπορούμε. Πάντως πολλά μπορεί να γίνουν σε επίπεδο και ιδιωτικών ναφών Υπάρχουν ενέφη ιδιωτικά εξαιρετικά διαχειριζόμενα και υπάρχουν και εφαρμογές οι οποίες δεν είναι πολύ επικίνδυνες και μπορεί να προχωρήσουν σωστά. Η κρυπτογράφηση σαν παράδειγμα είναι ένα καλό παράδειγμα μετακινεί κανείς το υλικό φυσικά με, με ε, κρυπτογραφημένο και αφού το μεταφέρει τότε μπορεί να το αναπτύξει και να το χρησιμοποιήσει. Οι κίνδυνοι δεν είναι τόσο μεγάλοι. Πάντως το πρόβλημα παραμένει. Είναι σοβαρό θέμα και πρέπει να αντιμετωπιστεί σωστά. The debate about whether or not this actually για τους κανόνες της FISA. Είναι κανόνες οι οποίοι είναι προβλέψεις υπερεδαφικές, εξωεδαφικές που ισχύουν για τον Αμερικανικό νόμο, καλύπτουν πολίτες εκτός Αμερικανικού εδάφου, μη Αμερικανούς πολίτες και είναι ρυθμίσεις οι οποίες στην ουσία είναι σε σύγκρουση με την Σύμβαση των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Η προσπάθεια την οποία κάνουμε εμείς είναι να προσπαθήσουμε εμείς να έχουμε να κάνουμε με επιχειρήσεις με αντιφατικές απαιτήσει από τις δημόσιες αρχές. Αν οι Αμερικανικές αρχές ζητούν δικαστικά, εν πάση περιπτώσει κάποια δεδομένα, νομίζουμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί μερικές φορές να έρχεται σε σύγκρουση με τα θεμελιώδη δικαιώματα όπως τα βλέπουμε στην Ευρώπη. Και γι' αυτό ακριβώς η προσπάθεια την οποία κάνουμε είναι πάρα πολύ σημαντική και επικίνδυνη για αυτούς οι οποίοι ε, λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους με, ε, ε, με νόμιμο τρόπο. Οι λύσεις που προτείνονται είναι ενδιαφέρουσες αλλά δεν είναι θα έλεγα ιδιαίτερα, δεν καλύπτουν τις ανάγκες που έχουμε για να λύσουμε τα προβλήματα. Από την συνάδελφο που εκπροσωπεί το Μπέκ. Κάποια από τα θέματα αυτά τα αντιμετωπίζουμε ήδη. Σε μία ανακοίνωση μπορεί να πει κανείς περιορισμένα πράγματα. Κάποιες οι προσπάθειες που κάνουμε σε επίπεδο συμβάσεων, σαν παράδειγμα, δεν εμπλέκουν άμεσα τους καταναλωτές, αλλά έχουν ενδιαφέρον και τα συζητάμε μαζί τους. και το θέμα της συνεργασίας ανάμεσα στις επιχειρήσεις γύρω από την διαδικασία αυτή. Πάντως είναι ένα αναδυόμενο φαινόμενο το νέφος, δεν έχει κανείς όλες τις απαντήσεις. Η φύση εν μια σύμβασης όταν κάποιος προτείνει μία λύση μέσω νέφους ή μία λύση λογισμικού γενικότερα, ε, οι απαντήσεις ποικίλουν, δεν μπορούμε να τα ενιοποιήσουμε όλα θα υπάρξουν κάποια κοινά στοιχεία και αυτό που απαιτείται είναι μεγαλύτερη, θα έλεγα, βασική διαφάνεια. Αυτή είναι η προσπάθεια την οποία κάνουμε στην Επιτροπή και ε, κατά τη διάρκεια του ενεστώτος έτους θα αναφερθούμε σε αυτά αναλυτικότερα. Γιατί τους όρους των συμβάσεων και την προστασία των καταναλωτών. Η συζήτηση είναι σημαντική. Αν διαβάσετε την ανακοίνωση προσεκτικά, αυτό που λέγεται είναι ότι έχουμε από τη μία την πρόταση για τον Ευρωπαϊκό Νόμο Πολίσεων, πιστεύουμε σε αυτόν, εμείς τον προτείναμε, και σε κάποιους τομείς άπτεται και των νεφών, των πληροφορικών νεφών. Και ανάλογα με το αποτέλεσμα των συζητήσεων για τον Ευρωπαϊκό Νόμο θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα δημιουργήσουμε μια ειδική ομάδα όμως να δει τα πράγματα και πέρα από αυτό. Αυτή είναι η διαδικασία στην οποία προσπαθούμε να εξοπλιστούμε, για την οποία προσπαθούμε να εξοπλιστούμε. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης είναι υπεύθυνη για τα θέματα αυτά έτσι ώστε ε, να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα σχετικά με τις ε, προτάσεις τις διακανονιστικές τις οποίες ε, θα προτείνουμε, τις οποίες θα καταθέσουμε. Τώρα για το ψηφιακό περιεχόμενο και το IPR δεν θα επιμείνω. Είπα ότι έτσι και αλλιώς σε κάποια φάση στο τέλος του χρόνου θα επανέλθουμε. Η χρήση ιδιωτικού και δημόσιου χώρου στο νέφος είναι κάτι το οποίο αποδεικνύεται χρήσιμο. Τώρα για την, ε, την δυνατότητα μεταφοράς ε, των δεδομένων. Είναι μια πολιτική πρόταση η οποία είναι συνδεδεμένη, καλύπτεται μάλλον από την πρόταση για την προστασία δεδομένων, θα καλύπτει και τις τεχνικές πλευρές και τις νομικές συμβατικές πλευρές. Ξέρω ότι η Μάργκο ασχολείται με αυτά. Στο έγγραφο λέγουμε ότι προσπαθούμε να διασφαλίσουμε τη διαλειτουργικότητα και την δυνατότητα μεταφοράς των δεδομένων με βάση τα συγκεκριμένα πρότυπα. Αυτή η προσπάθεια αφορά τον συντονισμό των προτύπων, δεν έχουμε καταλήξει ακόμα. Έχουμε μια ομάδα εργασίας που ασχολείται με τις τρεις αυτές τις, δυνατό... αυτές τις δυνατότητες. Να μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα του με σωστό τρόπο, με σωστή μορφή και με σωστό κόστος. Αυτά είναι θέματα που μας απασχολούν, αν και δεν έχουμε όπως είπα ακόμα καταλήξει και δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Η συζήτηση ήταν ενδιαφέρουσα, η συζήτηση για την ουδετερότητα του δικτύου είναι σωστή και δεν έχουμε επίσης μιλήσει ακόμα και για το λεγόμενο ευρύ φάσμα Αν χρησιμοποιεί κανείς ε, έτσι και αλλιώς ε, δημόσια δίκτυα, απαιτείται να έχει πάρα πολύ μεγάλο διαθέσιμο φάσμα για να υπάρχει και δυνατότητα ανταγωνισμού. Αυτά θα τα συζητήσουμε στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης τον μήνα Ιούνιο. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τη συζήτηση που ήταν ενδιαφέρουσα. Τώρα οι κατάλογοι έχουν, οι συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Η κυρία Τρότμαν, ευχαριστώ πολύ. Πιλάρ, έχω κάποιες επιπλέον ερωτήσεις. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές. Είναι συναρπαστικό το θέμα αυτό και αυτές οι παρουσιάσεις όλων των ζητημάτων και των προπτικών που μας προσφέρει το υπολογιστικό νέφος. Ταυτόχρονα είναι συναρπαστικά και αυτά τα ερωτήματα που γεννιόνται μέσα μας ως Ευρωπαίους. Πώς μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για επανεκκίνηση της ανάπτυξης, για επενδύσεις, για ανάκαμψη, για την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών μας, των, των διαφορών τομέων, πώς θα μπορέσουν να αποκτήσουν οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ενώ λόγω των ε, ρυθμίσεων που υπάρχουν ε, έχουμε δεσμευτεί ε, στο πλαίσιο μιας διεθνούς δραστηριότητας μπορεί να συναντήσουμε και συμφέροντα τα οποία δεν είναι επιτοπλίστων ευρωπαϊκά. Συμφωνούμε, πρέπει να αποφύγουμε τη ζούγκλα των προτύπων. Αλλά όταν μιλάμε για σύγκληση των προτύπων και υπάρχει το ενδεχόμενο αργότερα τα, να ανακαλύψουμε ότι αυτά τα πρότυπα ε, ωφελούν άλλους, μπορεί να μην κερδίσουμε το παιχνίδι. Ρωτάω λοιπόν πώς οι Κομισιόν καθώς και ο οργανισμός που μελέτα αυτά τα πρότυπα αντιδρούν, απαντούν σε αυτά τα ερωτήματα όσον αφορά την ασφάλεια. Θεμελιώδου σημασία ερώτημα. Συμφωνώ. Δεν μπορούμε απλά να πούμε ότι επειδή φυλάμε τα δεδομένα στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια είμαστε βέβαιοι για την ασφαλεία τους. Μόλις είπατε κύριε εκπρόσωπο της Κομισιόν ότι πρέπει να μπορέσουμε να αναπτύξουμε ένα δίκτυο ισχυρή ε, δυναμικότητας που να είναι ασφαλές με, και υψηλής χωρητικότητας. Ε, αυτή τη στιγμή το συνδέοντας την Ευρώπη δεν έχει τα κονδύλια. Θα πρέπει να βρούμε άλλα για αυτά τα δίκτυα. Επίσης, τίθε το ζήτημα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και το ζήτημα της προστασίας των δεδομένων. Ποιο είναι το καθεστώς το οποίο εφαρμόζεται. Υπάρχει σήμερα μια συγκεκριμένη απάντηση για τα δεδομένα που αποθηκεύονται από έναν Ευρωπαίο σε σερβερ στην Αμερική, για παράδειγμα, όταν αυτά έχουν προσωπικό χαρακτήρα. Όσον αφορά τι συμβάσει. άκουσα πολύ προσεκτικά τα όσα είπατε κυρία Πας Ξεκινήσατε με κάτι που εμάς στο Κοινοβούλιο μας φαίνεται θεμελιώδες, η εμπιστοσύνη. Αυτή τη στιγμή οι συμπολίτες μας μας υποβάλλουν ερωτήσεις και δεν έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη. Η εξοικονόμηση χρημάτων μπορεί να είναι ένα πιστικό επιχείρημα για να επιλέξει κανείς το υπολογιστικό νέφος είναι ενδιαφέρον, ε, κυρίως επειδή θα υπάρχουν διάφορες προσφορές, υπηρεσίες, αλλά μου φαίνεται ότι αυτό που είπατε στη σύστασή σας, οι συμβάσεις δεν μπορούν να αφορούν μόνο την πρόσβαση στο υπολογιστικό νέφος, αλλά και στην εφαρμογή του. Πώς συνδέεται αυτά τα δύο, πώς θα μπορέσουμε να το διατυπώσουμε σωστά. Αναφερθήκατε στην ουδετερότητα του δικτύου, εγώ πιστεύω ότι αυτή πρέπει να διαπνέει τις συμβάσεις. Όσον αφορά την πολυεδαφικότητα, σήμερα πιστεύω έχουμε ήδη εθνικά υπολογιστικά νέφη που είναι πιο γρήγορα από όσο μπορούμε να δώσουμε μια ευρωπαϊκή απάντηση. Πώς θα άρουμε αυτό το εμπόδιο, είναι σωστή αυτή η τακτική. Εσείς ε, αναφέρατε αυτή τη διαπίστωση, πώς θα αντιμετωπίσουμε τον ανταγωνισμό, πώς θα αποκτήσουμε μια πραγματική ενιαία αγορά, δεν έχουμε σήμερα μια αντίφαση. Η Κομισιόν προτείνει αφενός μια στρατηγική, για την άλλη έχουμε εθνικά υπολογιστικά ανέφη. Και όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τέλος, πολλοί συνάδελφοι, όπως και η Πιλαρ υποστηρίζουν ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θέλουμε να δώσουμε κίνητρα σε αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να επιλέξουν τις υπηρεσίες του υπολογιστικού νέφους. Για να οικοδοθεί καλύτερη στρατηγική λοιπόν χρειαζόμαστε μια παράθεση των αναγκών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ώστε να μπορέσουμε να τους προσφέρουμε αποδοτικές υπηρεσίες. Έχουμε δύο τύπους καταναλωτών, τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις. Οι ανάγκες τους δεν είναι απαραίτητα οι ίδιες. Αυτό πιστεύω είναι ένα στοιχείο στο οποίο θα πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα ώστε να οικοδομηθεί και αυτή η εμπιστοσύνη μεταξύ των επιχειρήσεων και να υπάρξει μια ανταπόκριση όσον αφορά τη δημιουργία δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων. Μήπω είναι απαραίτητο, τελευταία μου ερώτηση, να αναλύσουμε τι εφαρμογέ που ήδη χρησιμοποιούνται και να κάνουμε έναν απολογισμό ώστε ενδεχομένω να βελτιώσουμε την προτινόμενη στρατηγική και να την τροποποιήσουμε στα σημεία όπου είναι απαραίτητο. Είπατε κάποια στιγμή ότι ίσως ο κανονισμός ε, να μην είναι απαραίτητα το καλύτερο εργαλείο. Νομίζω κάποια στιγμή μιλήσατε για οδηγία επίσης. Έχουμε εδώ τα στρατηγικές πτυχές, αλλά έχουμε και τις πτυχές των νομικών ε, μέσων. Ζητώ συγγνώμη, είναι πολλές ερωτήσεις αυτές, ε, αλλά ε, πιστεύω ότι είναι σημαντικές και είναι και σημαντικές και για μένα ως και για την ομάδα μου. Ευχαριστούμε πολύ, ο κ. Τσανόφσκι. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι παρουσιάσεις σας. Και καλό θα ήταν αν μπορούσαμε να διαβιβάσουμε αυτές τις παρουσιάσεις και σε ένα πιο ευρύ φόρουμ. Είμαι πεπισμένος απόλυτα ότι στο, στον τομέα του κυβερνοχώρου πάντα είμαστε πίσω από τις εξελίξεις. Οι πολίτες δεν είναι προετοιμασμένοι. Έχουν περάσει στην καθημερινή χρήση πλέον τα smartphones, είναι ευρέως διαδεδομένα. Ενώ στην ουσία δεν έχει επακριβώς οριστεί τι γίνεται με τα προσωπικά δεδομένα αυτά. Και θα ήθελα λοιπόν να θέσω ένα φιλοσοφικό κάπως ερώτημα. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να αρθούν όντως τα εμπόδια τα οποία εμποδίζουν τις νέες τεχνολογίες να αναπτυχθούν όπως τα έπρεπε. Γιατί αυτό θα είχε μεγάλο όφελος. Από την άλλη πλευρά είναι δύσκολο να μειώσουμε το επίπεδο της νομικής προστασίας. Είμαστε σε θέση να αγγιηθούμε προστασία από όλους τους κινδύνους. Δεν θα πρέπει κανείς να αποδεχτεί σε ένα βαθμό το γεγονός ότι υπάρχει κάποιο ρίσκο, κάποιος κίνδυνος όταν διαθέτει τα δεδομένα του. Δεν πιστεύω ότι η προστασία θα μπορεί να είναι ποτέ απόλυτη. Ακόμα ε, όταν υπάρχει κωδικοποίηση, όταν υπάρχουν ε, διατάξεις ασφαλείας. Ποτέ δεν υπάρχει απόλυτη ασφάλεια και όσο πιο πολλές ε, τόσο πιο πολλά επίπεδα ασφάλειας προστίθενται, τόσο πιο ακριβές είναι αυτές οι υπηρεσίες. Και τελικά, είμαστε αντιμέτωποι με μια τεράστια πρόκληση. Και γι' αυτό λοιπόν θέλω να θέσω το εξή ερώτημα. Κατά πόσο στα πλαίσια της συζήτησή μας έχουμε αμελήσει μία πτυχή του θέματος. Αντιλαμβανόμαστε ποια κίνδυνοι υπάρχουν. Δεν έχει να κάνει αυτό με την ε, εμπιστοσύνη. Γνωρίζοντας ποιοι είναι οι κίνδυνοι οι οποίοι ε, υπάρχουν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ασφαλώς ε, θέλουμε να υπάρχει η κατάλληλη προστασία, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί και τέτοια προσέγγιση να ακολουθήσουμε. Εγώ είμαι ειδικό σε θέματα πληροφορικής και σε ό,τι αφορά θέματα που έχουν να κάνουν το διαδίκτυο, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί το περιεχόμενο ε, των κειμένων στο διαδίκτυο. Από πού και προέρχονται. Αυτό είναι ένας κίνδυνος τον οποίο λαμβάνω υπόψη. σε ό,τι αφορά για παράδειγμα συναλλαγές στο ίντερνετ. Αποδέχομαι τον κίνδυνο για παράδειγμα να χάσω τα χρήματά μου. Ξέρω όμω ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Ξέρω ποιοι είναι και οι κίνδυνοι όταν βγαίνω στον δρόμο και οδηγώ. Νομίζω λοιπόν ότι ο κόσμο θα πρέπει να αντιληφθεί του κινδύνου τη ψηφιοποίηση. Να μην δημιουργούμε την εντύπωση ότι με κάποιες δικλείδες ασφαλείας ε, μπορούμε να παρέχουμε την απόλυτη ασφάλεια. Και η απόκριση σε κάθε, τέτοια, σε κάθε τέτοιο κίνδυνο θα πρέπει να είναι εξατομικευμένη. Φυσικά υπάρχουν και κάποιοι κοινωνικοί ευθύνοι, αλλά είναι σημαντικό ο καθένας, το κάθε άτομο αντιλαμβάνεται τους κινδύνους. Να μην δίνουμε προπαντός την ε, εντύπωση ότι η κοινωνία προστατεύει το άτομο σε όλες τις πτυχές. Γιατί είναι πάρα πολύ περίπλοκο το ζήτημα αυτό, το ζήτημα του υπολογιστικού νέφους και δεν είμαστε καθόλου προετοιμασμένοι, σε καμία περίπτωση δεν είμαστε προετοιμασμένοι. Αυτό ήθελα να το θέσω ως φιλοσοφική σκέψη. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί, να δείξουμε ανοιχτό χαρακτήρα σε ό,τι αφορά την άρση των ε, τεχνολογικών εμποδίων. Επίσης θα πρέπει να προβούμε σε συμφωνίες με τρίτες χώρες. Θα πρέπει να υπάρχουν σχετικές πρωτοβουλίες, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τονίσουμε και την ευθύνη του ατόμου, γιατί ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι περίπλοκος, ανασφαλής, αβέβαιος. Και αυτά που ζούμε σήμερα τα βλέπαμε σε ταινίε επιστημονική φαντασία όταν ήμασταν μικροί. Δεν θα υπάρξει ποτέ το απόλυτα ασφαλέ νομικό πλαίσιο. Υπάρχουν κίνδυνοι. Και κάθε άτομο θα πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη. Δεν υπάρχει 100% προστασία. Και συγγνώμη αν μακρηγόρησε και αν μίλησα φιλοσοφικά μάλλον. Well, I think uh, it's all from uh, my colleagues uh, Αυτά από τους συναδέλφους. Τώρα μπορείτε να δώσετε κάποιες απαντήσεις αν θέλετε ή να σχολιάσετε αυτές τις δύο ενδιαφέρουσες ερωτήσεις από εντελώς διαφορετικές επόψεις. όλοι σας μπορείτε αν θέλετε να σχολιάσετε και να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από τους καταναλωτές. Ευχαριστώ για τα ενδιαφέροντα σχόλια και τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Θα ξεκινήσω με τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αναφέρθηκε σε αρκετά θέματα. Φυσικά λαμβάνουμε υπόψη μας ότι έχουν υπάρξει μέτρα σε σχέση με την τυποποίηση στον τομέα της δυνατότητας μεταφοράς δεδομένων, φορητότητας. the on the innovation, on the η καινοτομία θα επηρεάσει πάρα πολύ τις επιχειρηματικές δυναμικές, αλλά παρόλα αυτά δεν έχουμε δείγματα τα οποία να μας καθησυχάζουν σε σχέση με το βάρος, με τη σημασία που δίνεται έτσι ώστε να καταστήσετε το υπολογιστικό νέφος τμήμα, θα έλεγα, των δυνατοτήτων. Σχετικά τώρα με τα θέματα των όρων των συμβατικών, Υπάρχουν ε, δυνατότητες εδώ, υπάρχουν προβλήματα. Πρέπει να αναφερθώ σε αυτά τα οποία είπατε στη στρατηγική σας και δεν υπάρχουν αναφορές πέραν του Ευρωπαϊκού Νόμου Πολίσεων και κάποιων άλλων δυνατοτήτων κατ' επιλογή. Λέτε ότι θα πρέπει πριν από το και τους όρους έτσι ώστε οι καταναλωτές, η βιομηχανία και οι ομάδες εμπειρογνωμόνων να μπορέσουν να συνδυάσουν τις προσπάθειές τους και στα πλαίσια αυτής της εθελοντικής προσπάθειας να λυθούν και τα θέματα του υπολογιστικού νέφους που είναι παράλληλα με τα θέματα που θέτει ο Ευρωπαϊκός Νόμος Πολίσεων δεν είναι ιδιαίτερα ξεκάθαρη η σύνταξη αυτή, θα άκουσα με χαρά ότι θα επανέλθετε. Για τα σχόλια της κυρίας Τροτμάν και τις ερωτήσεις της, πολύ ενδιαφέρουσες, για τα θέματα των συμβάσεων, των όρων των συμβάσεων, πώς μπορεί να συνδυάσει κανείς τα θέματα της πρόσβασης με το περιεχόμενο και πώς μπορεί να κάνει σωστές επαφές. Το θέμα είναι τι μπορεί να συμπεριλάβει κανείς σε, ένα, σε μια σύμβαση με τους καταναλωτές. Ποια σύμβαση είναι δίκαιη και ισορροπημένη. Δεν έχουμε νομοθετικές ρυθμίσεις επακριβής για τον συγκεκριμένο τομέα. Γιατί και το υπολογιστικό νέφος και άλλες ψηφιακές υπηρεσίες θέτουν ξεχωριστά προβλήματα. Έχουμε μία θα έλεγα οδηγία η οποία αναφέρεται στις δίκες, ε, ε, στους δίκαιους όρους του συμβάσεις, στις συμβάσεις, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα για τα καταναλωτή να γνωρίζει και δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση ακόμα και για τα θέματα προσφυγής στη δικαιοδοσία της δικαιοσύνης. Δεν υπάρχουν ε, δεσμευτικές ρυθμίσεις για όλους και όχι μόνο εθελοντικές ρυθμίσεις όχι απλά να λέμε δηλαδή στον επιχειρηματικό κόσμο, αν τυχόν σας ενδιαφέρει και αν θέλετε μπορείτε να προχωρήσετε ε, σε ε, κάποιες ρυθμίσεις δίκαιες για όλους. για τα εθνικά νέφη, αν είναι σε αντίφαση με το ευρωπαϊκό νέφος. Καλή η παρατήρησή σας. Ξανά σε αυτό που είπα, ότι το βασικό εμπόδιο για μια ενιαία ψηφιακή αγορά είναι η πνευματική ιδιοκτησία. Εξορισμού το θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσει πλήρως τις ανάγκες των καταναλωτών, γιατί υπάρχουν υπηρεσίες στις οποίες έχει κανείς πρόσβαση από μία κάποια χώρα κάθε φορά και για τις άλλες χώρες απαιτείται ειδική αδειοδότηση κτλ. Ελπίζω να απάντησα στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Υπάρχουν σχόλια, θα πρέπει να είμαστε σύντομοι γιατί θα πρέπει να κλείσουμε σε λίγο. Θα είμαι πολύ σύντομος, θα ήθελα απλά να κάνω μερικές παρατηρήσεις. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλό που ο κύριος Ντουκατέλα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθεσε πολλά στοιχεία στη συζήτηση για αυτό το ζήτημα που ανέφερα εγώ και θα ήθελα να πω ότι είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που βλέπω ότι γίνεται μια σοβαρή συζήτηση για όλα αυτά τα ζητήματα και ότι γίνεται μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα και να εξευρεθούν λύσεις. Έγινε κάποια αναφορά στο να θεωρηθεί η ασφάλεια ως τεχνικό ζήτημα και συμφωνώ απόλυτα. Για πολλούς κινδύνους ασφαλείας ε, το να μεταφέρει κανείς τα δεδομένα σε πολύ ασφαλή ε, ε, υπολογιστικά νέφη υψηλής ποιότητας είναι Εξαιρετική ιδέα. Αλλά τώρα όσον αφορά την νόμιμη πρόσβαση και αυτό είναι ένα ζήτημα. Διότι και ιδιωτικά να είναι αυτά τα υπολογιστικά νέφη θα έχουν πίσω πόρτες και θα μπορούν να υποπέσουν σε παραβίαση πρόσβασης από κάποιες χώρες. Ας κάνουμε λοιπόν μια υπόθεση εδώ. Αν σχεδιάσουμε νομικές εξουσίες για αρχές επιβολής του νόμου και αρχές εθνικής ασφάλειας, θεωρείτε ότι είναι καλή ιδέα αυτές οι εξουσίες να εξαρτώνται από τον τόπο αποθήκευση των δεδομένων, θα είναι αρκετά εύκολη η παράκαμψή τους. Είναι πολύ λογικό τέτοιες εξουσίες ε, να είναι εδαφικές και όχι εκτός των εδαφών που αφορούν. Αυτή η ιδέα εδαφικότητας των δεδομένων αποτελεί ουσιαστικά το βασικό κίνητρο του κατά πόσο οι κυβερνήσεις, οι εθνικοί οργανισμοί θα έχουν έλεγχο αυτό το δεδομένο. Το ζήτημα είναι πολύ πιο ευρύ και θα πρέπει να κάνετε σχετική συζήτηση εδώ στο Κοινοβούλιο, διότι πολλά εδώ εξαρτώνται από αυτή την εδαφικότητα των δεδομένων και από το πού θα είναι αποθηκευμένα εκτός των εθνικών εφών. Αν οργανώσετε ας πούμε, ένα εθνικό ρεύμα, δεν σημαίνει ότι τα δεδομένα θα παραμείνουν στο Άμστερνταμ. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα και σίγουρα νομικά δεν είναι ο κατάλληλο τρόπο αυτό. Φυσικά ως πελάτης θέλετε να γνωρίζετε πού θα βρίσκονται τα δεδομένα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείτε να βασιστείτε σε αυτή την εδαφικότητα. Συχνά τα δεδομένα αυτά μπορεί να υπόκειται στη δικαιοδοσία πολλών χωρών και αυτό ουσιαστικά είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Για να απαντήσω για αυτό το ζήτημα του κινδύνου λοιπόν, της επικινδυνότητας, συμφωνώ απόλυτα. Είμαι κατά της ιδέας, δεν έχει νόημα να υπάρχει μια τέτοια κοινωνία ανευκινδύνου, αλλά πρέπει να συζητήσουμε τι κίνδυνοι είναι αποδεκτοί. Από την εμπειρία μου, όταν συζητάει κανείς με ανθρώπους και λέει μια ξένη κυβέρνηση μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα σας, ενώ εσείς θεωρείτε ότι είναι ασφαλή, οι άνθρωποι και οι κυβερνήσεις το θεωρούν απαράδεκτο. Και οι πολιτικοί. Από την αριστερά ή από τη δεξιά, οποιασδήποτε ιδεολογία θα το θεωρήσουν απαράδεκτο για πολύ καλούς λόγους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εμβαθύνουμε, να δούμε ποιους κινδύνους θεωρείται αποδεκτού και ποιους μη αποδεκτούς και γιατί είδους ασφάλεια μιλάμε σε αυτό το πλαίσιο. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ γρήγορη γιατί έκανε κάποιε συγκεκριμένε ερωτήσει η κυρία Τρότμαν για την τυποποίηση και πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας σε ένα παγκόσμιο σύστημα. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ερώτηση. Διότι ουσιαστικά αυτό που υπονοεί είναι ότι δεν υπάρχει ουδέτερη τυποποίηση, ανεξάρτητη τυποποίηση. Ή μάλλον οι εταιρείε έρχονται μια συγκεκριμένη ατζέντα στου οργανισμού τυποποίηση. Έτσι συμβαίνει, δεν είναι καλό ή κακό. Απλά έτσι έχουν τα πράγματα. αν θεωρείτε ότι η τεχνική επιρροχή είναι επαρκής ε, για να υλοποιεί η τεχνολογία σας το πρότυπο, αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε πάει σε αρκετές συναντήσεις περιτυποποίησης. Αυτό απεικονίζει απλά αυτά που συμβαίνουν στην αγορά. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα εμείς. Μια κρίσιμη μάζα οικοδομείται στην τυποποίηση και αυτό είναι ένα από του λόγου για του οποίου ε, οι εταιρείε έρχονται στο έτσι. Έχετε δίκιο λοιπόν. Μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα επειδή μιλάμε για παγκόσμια αγορά και πώ μπορεί να συμμετέχει κανεί διατηρώντα το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα και πώ μπορεί να διαβεβαιωθεί ότι αντλεί τα πλεονεκτήματα που θέλει να, να αποκομίσει. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει σχέδιο Β, δεν υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο. Διότι το εναλλακτικό σχέδιο είναι ότι δεν συμμετέχει για να μην χάσει το ανταγωνιστικό σου πλεονέκτημα και αυτό είναι κακό σχέδιο. Επίση, ε, άκουσα με ενδιαφέρον την ε, ερώτηση του Πολωνού βουλευτή, διότι ναι, αυτή η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο θέτει διάφορα ερωτήματα για τα οποία δεν έχουμε απαντήσεις. Κάτι που θεωρώ εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι η ιδιοκτησία στο υπολογιστικό νέφος και το πώς αυτό θα αλλάξει τη σχέση μας με τη μουσική, τα βιβλία, τα πάντα. Και εδώ βλέπουμε μόνο την κορυφή του παγόβουνου, μόνο την αρχή. Θυμάστε πριν από μερικά χρόνια δεν είχατε λογαριασμό στο Second Life, δεν ήσασταν κανένας, κανείς δεν μιλάει για το Second Life σήμερα. Κοιτάξτε τι συμβαίνει εδώ. Διότι εδώ ζούμε την πρώτη ζωή, το First Life. Γι' αυτό το λόγο. Δεν έχει κανεί λογαριασμό στο Second Life. Αυτά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Θα θέλετε να κάνετε κάποια σχόλια. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο γιατί απάντησαν και οι συνάδελφοι. Φυσικά το θέμα είναι οι επιχειρήσει, οι καταναλωτέ και η εμπιστοσύνη που έχουν. Επίση συμφωνώ απόλυτα με τον κ. Σουνάφσκι, τον Πολωνό βουλευτή, για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους που υπάρχουν. Αλλά είναι πολύ βασικό θέμα και το πώς μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο, με ποιους όρους, με ποιες συνθήκες. Πολύ βασικό. Και τώρα θα κλείσω με ένα τελικό σχόλιο, ακούγοντας αυτά που είπαμε σήμερα. Οι πιο πολλοί κίνδυνοι που αναφέρονται ε, είναι εγγενείς κίνδυνοι του συστήματος. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να αλλάξουμε, έτσι λειτουργεί το νέφος. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να ε, ελαστικοποιήσουμε αυτές τις αρνητικές ε, πτυχές. Και με, τον τρόπο, με ποιο τρόπο μπορούμε να το πετύχουμε αυτό, με μια ισχυρή ευρωπαϊκή ε, ένα ισχυρό ευρωπαϊκό κλάδο σε ό,τι αφορά την ψηφιοποίηση. Γιατί άλλο είναι να έχει κανεί τα στοιχεία, τα δεδομένα του στο Ισραήλ, και άλλο να τα έχει στην Ιταλία, για παράδειγμα. Αυτό που χρειαζόμαστε λοιπόν είναι μια ψηφιακή νέα αγορά. Μια αγορά που θα επιτρέψει την εξέλιξη μια ενιαία ευρωπαϊκή βιομηχανία και ίσω όρου λειτουργία για όλους εκτός Ευρώπης, προκειμένου να μην έχουμε μειονεκτήματα είτε σε ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων είτε σε ό,τι αφορά τους φόρους σε όλες τις πτυχές. Για να μην έχουμε δηλαδή ε, άλλες επιχειρήσεις που θα θέτουν σε κίνδυνο τις δικές μας επιχειρήσεις. Νομίζω ότι μια ισχυρή ευρωπαϊκή βιομηχανία, ένας ισχυρός, βιομηχαν... ένας ευρωπαϊκός κλάδος θα είναι το καθαριστικό στοιχείο. Τελευταία σχόλια, καταρρεκτικά σχόλια, θα μιλήσω τη γλώσσα μου, στα ισπανικά. Eh, Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους συζήτητες. Νομίζω ότι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα μας έδειξαν τι δυνατότητες υπάρχουν και μπορέσαμε να εμβαθύνουμε στο θέμα παρότι ο χρόνος ήταν σύντομος. Έχω την αίσθηση ότι το φαινόμενο αυτό είναι ένα παράδειγμα, ένα υπόδειγμα που έχει πολύ μεγάλη σημασία σε σχέση με τις επιπτώσεις της παγκοσμιότητας ε, που ζούμε. Όπως είπε και ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, είναι ένα αναδυόμενο φαινόμενο. Και όπως όλα τα αναδυόμενα φαινόμενα, είναι ένα φαινόμενο εν κατασκευή. Και σε επίπεδο τεχνολογίας ε, της πληροφορικής, η οποία εξελίσσεται με τρομερή ταχύτητα, και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν προσπαθούμε ε, να παγώσουμε και να παγιώσουμε κάποιες λύσεις ε, σε επίπεδο νομικό, σαν παράδειγμα το θέμα της ρύθμισης της νομικής της δραστηριότητας αυτής. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να καλύψει κανείς όλες τις ανάγκες γιατί τα πράγματα αλλάζουν συνεχώς. Είναι ένα εγκατασκευή μη στατικό φαινόμενο και παρουσιάζει ένα εξαιρετικό δυναμισμό. Παρ' όλα αυτά, η ισορροπία ανάμεσα στις απαντήσεις στα πραγματικά προβλήματα τα οποία πρέπει να δώσουμε, στα θέματα που άπτονται του δικαίου των συμβάσεων, στα δικαιώματα των καταναλωτών, στα ε, δικαιώματα και στις ανησυχίες των επιχειρήσεων, είναι σαφές ότι δεν θα πρέπει να περάσουμε σε μια διακανονιστική λύση η οποία είναι τελικού αποφασιστικού τύπου, αμετακίνητη η οποία δίνει εγγυήσει για τα πάντα όπως είπε ο συνάδελφος το Σενόφσκι, που δίνει να πιστεύουμε, που κάνει να πιστεύουμε ότι όλα μπορεί να επιληθούν σε μια δεδομένη στιγμή και ότι υπάρχει η απόλυτη ισορροπία. Όχι, το φαινόμενο είναι δυναμικό, το φαινόμενο είναι εγκατασκευή, το φαινόμενο είναι αναπτυσσόμενο και πρέπει να υπάρξουν οι δυνατότητες έβρεσης λύσης στα προβλήματα αυτά, προβλήματα τα οποία αποτελούν την πραγματικότητα. Αυτό είναι το κλειδί, αυτό είναι το πεδίο στο οποίο θα πρέπει μέσα σε αυτό το πλαίσιο και υπάρχει η ατομική ευθύνη, η οποία αποκτά μεγάλη σημασία και επαναλαμβάνω ότι η ατομική ευθύνη σε ένα ανοιχτό κόσμο είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι αντίστοιχα σε σύνολα κλειστά, σε σύνολα δικτατορικά, σε σύνολα αυταρχικά. Όπου εκεί δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί επιβάλλονται τα πράγματα στο άτομο αλλά παρόλα αυτά στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε σφαιρικά φαινόμενα και θα πρέπει να προτείνουμε και να βάλουμε στη σωστή θέση την έννοια της ατομικής ευθύνης. Έχει μεγάλη σημασία και σε φιλοσοφικό επίπεδο, αλλά πρέπει να βρούμε κάποιες απαντήσεις στα θέματα τα λειτουργικά, στα θέματα τα συμβατικά, στα θέματα τα νομικά κτλ μια, ένα επίπεδο ισορροπίας ψάχνουμε, αυτή είναι η αναζήτηση και αυτή είναι η ευθύνη την οποία πρέπει να έχουμε όλοι, όλοι οι τομείς, όλη η κοινωνία και η βιομηχανία και οι καταναλωτές. Αυτό είναι το συμπέρασμα λοιπόν στο οποίο καταλήγω στην παρούσα φάση, είναι μια φάση σε κίνηση για το Κοινοβούλιο και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε αν θέλετε κάποιες πλευρές να τις αναλύσουμε σε επίπεδο λεπτομέρειας και να καταλήξουμε στη στρατηγική που θέλει να μας παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία θα πρέπει να είναι μια καλή και έλογη πρόταση. Ευχαριστώ. Κλείσαμε λοιπόν την δημόσια αυτή ακρόαση για το υπολογιστικό νέφος, το cloud computing. Ευχαριστώ όλους τους εισηγητές και την κυρία Πιλάρ. Και περνάμε τώρα στο τελευταίο θέμα της ημερησίας διάταξης των εργασιών μας, αφού χαιρετήσουμε τους εισηγητές ομιλητές.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 θα καλέσω εδώ στη συνέχεια τον Διευθυντή Πολ Τίμερς. Στο μεταξύ ήθελα να σας να ανακοινώσω στην Επιτροπή το αποτέλεσμα της απόφασης των συντονιστών που ελήφθησαν χθε. Η ΙΤΡΕ αποφάσισε να οργανώσει μια συνάντηση για το θέμα της ενέργειας σε συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια και με τη Λιθουανία. Στη συνέχεια θα ζητηθεί εξουσιοδότηση για έκθεση πρωτοβουλίας για την Πράσινη Βιβλία και την Ενέργεια που ανέλαβε το ECR. Το ECR επίσης ανέλαβε μια γνωμοδότηση για το CCS και για τα FEE δίκτυα. Το ΕΛΚ ενημέρωση για τις μεγάλες επιχειρήσεις, το COP19 και τη βιομηχανία στο δομέα της άμυνας. Έχουμε ολοκληρώσει εδώ την ενημέρωση για τη χθεσινή συνάντηση συντονιστών και περνάμε στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Δίνουμε το λόγο για την παρουσίαση περί διευρωπαϊκών δικτύων επικοινωνιών στον διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Connect, Paul Timmers, για 10 λεπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σαρτόρια και ευχαριστούμε πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να επανέλθω εδώ με μια σύντομη παρουσίαση για την τροποποιημένη πρόταση για τη διευκόλυνση ε, συνδέοντα την Ευρώπη για τις τηλεπικοινωνίες και τις κατευθυντήριες γραμμές. Ε, είχα το σκοπό να σας δείξω κάποιες διαφάνειες, αλλά για να μην χάσουμε χρόνο θα ξεκινήσω ήδη. Περιγράφοντάς σας ε, κάποια πράγματα που ήδη γνωρίζετε πολλοί από εσάς. Όπως γνωρίζετε εδώ βρισκόμαστε στη διαδικασία να σας παράσχουμε μία τροποποιημένη πρόταση που είναι το αποτέλεσμα συζητήσεων ε, στο πλαίσιο των επαφών για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο όπου η τρέχουσα κατάσταση με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τη σχετική πρόταση μείωσης του προϋπολογισμού από 9,2 δις ε, κατά ε, δις σχεδόν και οι αντίστοιχε συζητήσει στην ε, σχετική επιτροπή του Κοινοβουλίου μα κατέδειξαν ότι χρειαζόταν να τροποποιήσουμε την πρόταση. Μιλάμε λοιπόν για μια κατάσταση όπου ξεκινάμε από μια αρχική πρόταση 9,2 δισεκατομμυρίων σε κάτι που προτείνεται να είναι 4,1 δισεκατομμύρια. Εκεί είχαμε σκόπο να δώσουμε 7, δις στις ευρωζωνικές υπηρεσίες και το υπόλοιπο για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Είμαστε πεπισμένοι ότι θα χρειαστεί εδώ να αντιμετωπιστεί η ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών ώστε να διευκολυνθεί και η ευρυζωνική υπηρεσία. Έτσι προτείναμε να μειωθεί ο αριθμός των ψηφιακών υπηρεσιών και των σχετικών υποδομών που θα είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση. Αυτό είναι το ένα στοιχείο και να περιοριστεί το ευρώ τη υποστήριξη στις υπηρεσίες ε, Αυτό μας έδωσε και την ευκαιρία να βεβαιωθούμε ότι η πρόταση θα είναι πιο απλή και ελπίζω ότι υπό αυτή την έννοια θα είναι και πιο συμπαγής, πιο εύκολο να την παρακολουθήσει κανείς. Δεύτερον, ελπίζουμε ότι θα αντικατοπτρίζει πολλές από τις τροπολογίες που προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήδη όσον αφορά ειδικότερα τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες. Ε, την αντιμετώπιση τη ουδετερότητας του δικτύου, τη επενδύση του ιδιωτικού τομέα και τη παρεμβάση από χρηματοδοτικά μέσα. Και θα αντικατοπτρίζει επίση τη συζητήση του Συμβουλίου τη διαγραφή συγκεκριμένων διατάξεων για κατεξοδότηση πράξη. Να σα πω πρώτα δύο λόγια παραπάνω, γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε η πρόταση εστιάζεται πλέον περισσότερο στι υποδομέ ψηφιακών υπηρεσιών. Και Χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να πω δύο λόγια παραπάνω για αυτέ, για να ανακεφαλαιώσω το θέμα για το οποίο μιλάμε, γιατί η ορολογία είναι λίγο δύσκολη. Οι υποδομέ ψηφιακών υπηρεσιών αποσκοπούν να παρέχουν σε όλη την Ευρώπη τη δυνατότητα για του πολίτε, τι επιχειρήσει, τι δημόσιε αρχέ να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίε αδιάκοπα, online. Για παραδείγμα, παροχή πρόσβαση σε αρχεία υγεία για τη συμμετοχή σε δημόσιε συμβάσει για την πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο παντός είδους υπηρεσίες. Πολλές από αυτές τις υπηρεσίες ε, στην πραγματικότητα οικοδομούνται με ε, οικοδομικούς λίθους θα λέγαμε, building blocks, ε, δηλαδή ας πούμε την αδιακόπη πρόσβαση στην ηλεκτρική ταυτοποίηση που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς σε πολλά περιβάλλοντα. Είναι λίγο τεχνικό αλλά είναι σημαντικό να καταλάβετε ότι πρέπει να δημιουργηθεί αυτό το σύνολο των building blocks και πάνω σε αυτό να δημιουργηθούν οι υπηρεσίες έτσι ώστε να δημιουργείται όλο και μεγαλύτερη προστέμενη αξία αυτή η ηλεκτρονική ταυτοποίηση και η σχετική πρόσβαση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ε, δημόσια συμβάση, για επίλυση διανέξεων online ή για την πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο. Αυτά τα μπλοκ λοιπόν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες περιπτώσεις και αποτελούν στοιχείο των ψηφιακών υπηρεσιών. Ένα τέτοιο παράδειγμα οικοδομήματος ε, φανταστείτε ηλεκτρονικές παραδόσεις. Ηλεκτρονική παράδοση, δηλαδή ηλεκτρονικών εγγράφων, πολύ σημαντικό ας πούμε για να συνταγογραφήσει ένας γιατρός φάρμακα από τη μια χώρα σε μια άλλη, κάποιος τουρίστρα ας πούμε από μια χώρα που επισκέπτει την Αυστρία, από την Ολλανδία μπορεί ξέρω, να λάβει τη συνταγή του από τον γιατρό του με ασφάλεια μέσω διαδικτύου. Αυτή είναι η ηλεκτρονική παράδοση και η ηλεκτρονική υγεία μια πλήρης υπηρεσία που θα χρησιμοποιεί αυτό το block του e-delivery της ηλεκτρονικής παράδοσης γιατί η ίδια ασφάλιση παράδοση ε, γράφου μπορεί να γίνει επίσης και σε περίπτωση που μια ε, εταιρεία κάνει πρόταση, κάνει κάποια πρόταση για κάποια δημοσία σύμβαση. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε αυτά τα τουβλάκια ως ε, τουβλάκια πολλαπλών χρήσεων και που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλές υπηρεσίες. Πώς λειτουργούν οι ψηφιακές υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ευρώπη, μπορεί να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες σε όλες τις χώρες. Για παράδειγμα, στις ηλεκτρονικές δημοσίες ω ως εταιρεία έχετε το δικαίωμα να κάνετε μια προσφορά για μια δημοσία σύμβαση σε μια άλλη χώρα, μπορείτε να το κάνετε για πρόσβαση σε ηλεκτρικά αρχεία υγείας, για παράδειγμα εδώ στο το παράδειγμα τουρίστα. Λειτουργούν λοιπόν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πρόκειται για ένα πραγματικό διευρωπαϊκό τρόπο ανταλλαγή πληροφοριών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Υπάρχουν ψηφιακέ συνδέσει σε όλη την Ευρώπη, αλλά είναι πιο πυκνέ από του αυτοκινητόδρομου, διότι παρέχουν μια σειρά από υπηρεσίε στου ε, χρήστε. Για παράδειγμα, η κόρη μου μπορεί να εγγραφεί έτσι σε ένα πανεπιστήμιο σε μια άλλη χώρα. Οι, Οι υποδομέ λοιπόν ψηφιακών υπηρεσιών αποτελούνται από αυτά τα τουβλάκια Μιλάμε για τη διατηρητικότητα των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, ηλεκτρονικέ υπογραφέ εγγράφων, ηλεκτρονική παράδοση που μόλι ανέφερα, αυτόματη μετάφραση, θα μπορούσε να είναι ένα άλλο καλό παράδειγμα. Και οι υπηρεσίε που έχουν ιδιαίτερη αξία από πρακτική άποψη είναι υπηρεσίε μεταξύ κυβερνήσεων, κυβερνήσεων προ πολίτε, ηλεκτρονικέ δημόσιε συμβάσει, ηλεκτρονική υγεία, πρόσβαση σε ελεύθερης χρήσης δεδομένα, κινητικότητα επιχειρήσεων, πρόσβαση σε πολιτιστική κληρονομιά και ασφαλέστερο διαδίκτυο για τα παιδιά, καθώς και άλλες διασυνοριακές υπηρεσίες. Χαίρομαι που επαναρχόμαστε σε αυτό. Όπως βλέπετε στην εικόνα, ανεχτέ μια γέφυρα όπως η ψηφιακή υπηρεσία. Η γέφυρα αυτή οικοδομείται με τα τουβλάκια αυτά, τα πολλαπλών χρήσεων. Εδώ βλέπετε έναν πίνακα ένα σχεδιάγραμμα που βλέπετε στους καθούς άξονες, έχετε τα τουβλάκια, την ηλεκτρονική υπογραφή, την ηλεκτρονική παράδοση, την ηλεκτρονική ταυτοποίηση, την ηλεκτρονική τιμολόγηση και την υποστήριξη ασφαλείας και στην οριζόντια πλευρά βλέπετε τις υπηρεσίες, τις ψηφιακές υπηρεσίες που χρησιμοποιούν αυτά τα τουβλάκια. Δημόσια συμβάσεις, κινητικότητα επιχειρήσεων κτλ. Έτσι οικοδομείται ένα σύστημα ψηφιακών ευκαιριών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τώρα, οι αναθεωρημένε κατευθυντήριε ε, γραμμέ του ΣΕΤ λένε ότι κατά προτεραιότητα αυτά τα τοβλάκια θα πρέπει να υποστηρίζονται μόνο όταν είναι έτοιμα, όχι υπό την παρουσία του μορφή, οι ψηφιακέ υπηρεσίε που χρησιμοποιούν αυτά τα τουβλάκια και που είναι απαραίτητε για την υλοποίηση συγκεκριμένων νομοθεσιών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλων ψηφιακών υπηρεσιών. Οι απαιτήσει, και αυτό είναι σημαντικό να τονιστεί, ότι αυτό που θα υποστηρίζεται πρέπει να είναι όριμο δεν πρόκειται εδώ για ένα πρόγραμμα έρευνα και ανάπτυξη. Μιλάμε για εφαρμογή πραγμάτων που πραγματικά λειτουργούν στην πρακτική. Ήδη χρησιμοποιείτε πολλά από αυτά στα κινητά σα τηλέφωνα και ελπίζω να τα χρησιμοποιείτε πολύ. Συνεπώ αυτά πράγματα πρέπει να λειτουργούν σωστά καθημερινά σε 24 ώρε το 24 ώρο, 7 ημέρε τη βδομάδα. Πρέπει λοιπόν να έχει οριμάσει ω τεχνολογία και να βασίζεται σε ένα μακροπρόθεσμο οικονομικό επιχειρηματικό σχέδιο. Πώς το λειτουργεί κανείς αυτό πρέπει να βασιστεί μακροπρόθεσμα σε ένα οικονομικό σχέδιο, διότι αυτέ οι υπηρεσίε δεν θα υπάρχουν μόνο μέχρι το 2020 στο πλαίσιο τη διευκόλυνση ιδιότητα στην Ευρώπη, θα διαρκέσουν περισσότερο, ελπίζουμε. Κάποιε μπορεί να χρειαστούν δημόσιε επενδύσει, χρηματοδότηση, αλλά μπορεί και να δημιουργήσουν έσοδα, διότι χρησιμοποιούνται πραγματικά. Το ε, μοντέλο λοιπόν χρηματοδότηση μπορεί να μεταβάλλεται μέσα στον χρόνο, ξεκινώντα από τη διευκόλυνση το συνδέοντα την Ευρώπη και τη σχετική χρηματοδότηση, η οποία θα εξαλειφθεί σταδιακά, ίσως όχι για όλε αλλά για κάποιε από αυτέ. Αυτό θα γίνεται κατά περίπτωση τώρα. Το, το κομμάτι των ευρυζωνικών υπηρεσιών θα υποφεληθεί και το ICT θα αποτελέσει πιθανότητα το τέταρτο θέμα συγκέντρωση στο πλαίσιο του ΕΣΕΦ και ορισμένα κρατημέλη θα αναζητήσουν τρόπου για να αυξήσουν την αξιοποίηση και την οικονομική αποδοτικότητα των δαπανών του σε ευρυζωνικέ υπηρεσίε η ψηφιακή χρηματοδότηση για τις ευρυγιζονικές υπηρεσίες ε, στο πλαίσιο του ΣΕΦ προτείνουμε να περιοριστεί στο seed funding, ε, δηλαδή μιλάμε για χρηματοπιστωτικά εργαλεία στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτό συζητήθηκε σε μια συνέντευξη που είχαμε στο Στρασβούργο πρόσφατα και είδαμε ότι έχουμε την ε, η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Εδώ μπορούμε να επιφεληθούμε από την εμπειρία και την προγνωμοσύνη της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με αποτέλεσμα απευθείας χρηματοδότηση μιας ε, σειράς υποδειγματικών έργων που θα βοηθήσουν να προσελκύσουμε ε, επιμέρους συμβολές από τα κράτη-μέλη και ιδιωτικές επενδύσεις από επενδυτές που αναζητούν ευκαιρίες στην Ευρώπη. Και εδώ πιστεύουμε ότι θα μπορέσουν να έρθουν πολύ σωστά αποτελέσματα χάρη σε μια μικρή χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά όργανα. Η πρόσβαση λοιπόν είναι ότι θα συμβάλλει το ΣΥΕΦ το στην Ευρώπη για τις μεταφορές στην ενέργεια, τις ψηφιακές υπηρεσίες και θελοντικές συμβουλές, για παράδειγμα από τα κράτη-μέλη, από τα δικά τους ε, από τη δική τους συμβουλή, από το δικό τους μερίδιο στο ESIF, ε, στο Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία. Το, η διευκόλυνση σύνδεση στην Ευρώπη συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και με πιθανή εμπλοκή άλλων κάποιων τραπεζών για προώθηση και θα βοηθήσει να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο στον τομέα των ευρυζωνικών υπηρεσιών. Έχουμε λάβει υπόψη πολλά από τα αιτήματα τροπολογιών που έχουν προελθεί από το Κοινοβούλιο στον τομέα των ευρυζωνικών υπηρεσιών. Ελπίζω να μην μίλησα υπερβολικά πολύ και έχετε το λόγο κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο Τοσενόφσκι, ο οποίος είναι εισηγητής για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομος γίνεται. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι. Εμείς πήραμε το τροποποιημένο κείμενο πρόσφατα και πρέπει να συζητηθεί το ταχύτερο δυνατόν γιατί κατανοούμε το σύνολο αυτού του προβλήματος. Και γι' αυτό τον Ιούλιο θα πρέπει να υπάρξει το τελικό κείμενο, το διορθωμένο. Το αρχικό κείμενο το είχαμε ήδη υιοθετήσει στην Επιτροπή μας τον προηγούμενο Νοέμβριο. Εν τω μεταξύ υπήρξαν ορισμένες λεπτομέρειες, περάσαμε από τα 9,2, περάσαμε στο 1 δις, από 9,2 δις. Και αυτό φυσικά επηρεάζει ιδιαίτερα το τροποποιημένο πρόγραμμα. Το έχουμε συζητήσει επανειλημμένα. Πάντως από τον προηγούμενο Νοέμβριο συνάντησα επανειλημμένα την Επίτροπο και τους συναδέλφους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την Επιτροπή, συγγνώμη. Στο Στρασβούργο είχαμε τη δυνατότητα να συναντηθούμε με την Ιδία την Επίτροπο και τους εκπροσώπους των υπηρεσιών της, το σκιώδης εισηγητές. Όλοι έχουμε εμπλακεί στις συζητήσεις αυτές. Προσπάθειές μας είναι να προσπαθήσουμε να σεβαστούμε την χρονική προθεσμία που έχουμε που είναι πάρα πολύ ε, συγκεκριμένη και απαιτητική θα έλεγα, να συζητήσουμε λοιπόν αυτό το κείμενο και να αντιδράσουμε στις τροπολογίες έχουν κατατεθεί έτσι ώστε να τις εντάξουμε στην διορθωμένη, ε, στην διορθωμένη έκθεση. Νομίζω ότι η διαδικασία θα πάει καλά γιατί έχουμε ήδη περάσει πολύ χρόνο συζητώντας, συζητώντας συγγνώμη, τα προβλήματα αυτά. Ελπίζω να καταλήξουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Υπήρχε ένα θέμα σχετικά με την παρουσίαση την οποία μόλις ε, ακούσαμε για τις συστημικές υπηρεσίες ε, και ε, το ευρύ φάσμα, την ευρυζωνικότητα. Εδώ τίθεται λοιπόν η ιδέα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι σκοπεύει να κάνει γύρω από το θέμα αυτό. Η παρουσίαση που κάνατε ήταν ενδιαφέρουσα αλλά πολύ σύντομη και δεν είμαι βέβαιος ότι καταλάβαμε πάρα πολύ καλά αυτά που είπατε για την ευρυζωνικότητα. Ευχαριστώ συνάδελφο Ντερκαστήγιο. Ευχαριστώ. Έχω ένα, μια δήλωση από τον συνάδελφο Χόκμαρκ, ε, πρόεδρε, που είναι ο σκιώτης του ΕΛΚ. διαβάσω. Η ψηφιακή οικονομία χρησιμοποιείται κυρίως για ανάπτυξη. Για να αναπτύξουμε το δυναμικό της, λοιπόν, θα πρέπει να ακολουθήσουμε συγκεκριμένα μέτρα μετά από τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το EMFF ε, στις αρχές του έτους ο, τα κονδύλια για την ευρυζωνικότητα και τις ψηφιακές υπηρεσίες περικόπηκε ε, δραστικά από 9 δισεκατομμύρια σε 1 δισεκατομμύρια για την αξιοποίηση των ευκαιριών του ευρυζωνικότητας. Δεν ε, είναι αυτός ο σωστός τρόπος όμως. Αν θέλουμε να εξέλθουμε από την οικονομική κρίση, είναι σημαντικό να τεθούν οι σωστές προτεραιότητες στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. αλλά οι περικοπές σε τομείς όπως η ευρυζωνικότητα δεν είναι η λύση. αντιθέτω. είναι αντιπαραγωγικό. Δεδομένη της οικονομικής κατάστασης, είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να αντισταθμίσουμε αυτές τις οικονομικές ε, περικοπές, επιτρέποντας ε, χρηματοδότηση από τα διευθυντικά ταμεία. Ας χρησιμοποιήσουμε καλύτερα λοιπόν τα ταμεία αυτά για να επενδύσουμε στο μέλλον αντί να διατηρήσουμε παλές δομές. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το η Επιτροπή η βιομηχανία ε, ψήφισε τις αρχικές κατευθυντήριες γραμμές στο περσινό έτος, λάβαμε υποστήριξη για πιο φιλόδοξους στόχους και πιο αυστηρά κριτήρια για τις επενδύσεις στην ευρυζωνικότητα. διασφαλίζοντας ε, ότι θα υπήρχαμε 100 GB στη Συνήπεθρο και περισσότερα στις αστικές περιοχές. Η Ήπεθρο δεν θα πρέπει να μείνει πίσω. Θα πρέπει να είναι εξίσου διασυνδεδεμένη όπως και όλα τα άλλα μέρη της Ευρώπη. Είναι φιλόδοξα τα κριτήρια αυτά που θα πρέπει να επιβληθούν για την Ήπεθρο για να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα. Σημειώνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει συμπεριλάβει τους στόχους αυτούς στις αναθαρρυμένες προτάσεις της. Ωστόσο, θα συνεχίσουμε να προωθούμε αυτούς τους φιλοδοξούς στόχους και προσβλέπω στις μελλοντικές συζητήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ τη συνάδελφα Καστήλιο και Κρέφμαν. Κύριε Κρότσμαν, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καινούργια πρόταση, να τη συγχαρώ κιόλα. Πρέπει φυσικά να εξετάσουμε τι λεπτομέρειε του νέου κειμένου, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο βήμα προς σωστή κατεύθυνση. Θέτει σωστά, σωστό επίκεντρο σε ό,τι αφορά τα κονδύλια, σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα έργα. Θεωρώ ότι προσθέτει ε, ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Ήμουν αρκετά σκεπτικιστικό στην αρχή ε, σε ό,τι αφορά την ευρυζωνικότητα. Θεωρούσα ότι τα κράτη-μέλη έπρεπε να δραστηριοποιηθούν γιατί τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ πολλοί από τους συμμετέχοντες της αγοράς θεωρούν ότι είναι ένα ελάχιστο ποσό σταγόνα στον ωκεανό. Και φυσικά το θέμα είναι μήπως τα χρήματα αυτά θα έπρεπε να έχουν δαπανηθεί σε άλλο τομέα. Η νέα πρόταση θέτει το επίκεντρο στις υποδομές για τις ψηφιακές υπηρεσίες και απλοποιείται. Τα φλέγοντα ερωτήματα έχουν να κάνουν με το νομοθετικό έργο της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ηλεκτρονικές υπογραφές ε, και τα ψηφιακά αυτά προϊόντα έχουν τεράστιο δυναμικό. Χρειάζονται λοιπόν τα έργα αυτά προκειμένου η νομοθεσία που θέλουμε να έχει εφαρμοστεί μέχρι τη τέλη της θητείας να εφαρμοστεί όντως. Και σημαντικό είναι να συνδεθούν τα εθνικά μητρώα και έτσι θα μπορέσουμε να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για την πρόθεση της οικονομίας. Χαίρομαι που το PNR δεν έγινε θύμα. Τα υπόλοιπα τα έργα φυσικά θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν με μακροπρόθεσμο ορίζοντα για να, χρειάζεται, για να υπάρχει η ασφάλεια σχεδιασμού χωρίς περικοπές. Τέλος, θα ήθελα να μιλήσω για το θέμα του διαδικτύου. Κάποια θέματα, κάποια έργα είναι αφιλεγόμενα. Αλλά δεν θα ήθελα να ξισωθεί αυτό σε ό,τι αφορά τις ε, ικανότητες ε, συμμετοχής στον τύπο γονέων και παιδιών. Μας ε, φτάνουν οι ανησυχίες των γονέων που μας αναφέρουν τα των περικοπών για τη σχετική πολιτική σε ό,τι αφορά το Connecting Europe Facility. Φαίνεται ότι αποτελεί ένα βασικό μέτρο για το κατά πόσο τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τέτοια ζητήματα. Αυτό δεν είναι σαφές. Γι' αυτό λοιπόν ρωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορούμε να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε και να χρηματοβούμε τα προηγούμενα έργα που ήδη υφίστανται ή θα πρέπει να συγχρηματοδοτούν και τα κρατη Και αν ναι, θα το κάνουν. Και επαναλαμβάνω πολλά επιδοτούμε και προωθούμε στην Ευρώπη, αλλά όταν τίθεται θέμα ανθρώπου, ο άνθρωπος ε, καταλαβαίνει ποια είναι η προστιθόμενη αξία της Ευρώπης. Και είναι κρίμα, γιατί δεν πρόκειται για μεγάλα ποσά. Ιδιαιτέρως αυτά τα προγράμματα που πραγματικά αγγίζουν τον πολίτη τότε δεν θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν σε αυτά τα προγράμματα, σε αυτά τα έργα, να κάνουμε περικοπές. Ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε περικοπές, αλλά όχι να τα καταργήσουμε εντελώς. Ίσως να εξετάσουμε την δυνατότητα της χρηματοδότησης. Αλλά είναι πραγματικά πάρα πολύ κρίμα όταν ο κόσμος βλέπει ότι κάτι κάνει η Ευρώπη για τον πολίτη, ξαφνικά να σταματάνε τα προγράμματα και να λέει η Ευρώπη ότι αν δεν μας ενδιαφέρουν πλέον τα προγράμματα αυτά. Πολλά είναι τα αμφιλεγόμενα προγράμματα και μάλιστα που, ε, στα οποία δαπανούμε πάρα πολλά κονδύλια. Αλλά ίσως λοιπόν αυτά τα προγράμματα που έχουν συγκεκριμένο αντίκτυπο θα πρέπει να τα κρατήσουμε. Ωραία, ευχαριστούμε και ως συνάδελφος ε, Ήθελα να προσθέσει κάτι ο συνάδελφος από την Κομισιόν. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για τα σχόλιά σας και τη θετική σας προσέγγιση για ταχεία προώθηση αυτής της ατζέντα. Θεωρούμε ότι και εμείς, και εμείς θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά σπουδαία και όπως είπε και ο κ. Στουσανόφσκι μπορεί να υποφεληθεί από τη στενή συνεργασία που είχαμε μέχρι στιγμής καθώς και από τις εντατικές ε, προετοιμασίες που έχουν λάβει χώρα. Μέσω όλων αυτών πιστεύω κατανοήσαμε καλύτερα τι θέλουμε να επιτύχουμε, ποια είναι η φύση αυτών των έργων κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και το πόσο είναι εφικτά. Το σαφές μήνυμα που δίδει, δόθηκε είναι ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε σε έναν κόσμο όπως είχαμε προβλέψει Έχουμε 9 δισεκατομμύρια ανθρώπους και ο τρόπος ε, με τον οποίο αγγίζουμε τις ευκαιρίες του ευρυζωνικού δικτύου είναι διαφορετικές και το γεγονός ότι το ICT μπορεί να γίνει μια τέταρτη προτεραιότητα και το ότι έχουμε μια θετική εντύπωση για το πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα χρηματοδοτικά μέσα μαζί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πιστεύουμε ότι παρέχει σημαντικές ευκαιρίες για να τηρήσουμε, να εκπληρώσουμε τις φιλοδοξίες του ευρυζωνικών υπηρεσιών. Από αυτή την άποψη επίσης ε, θα ήθελα να επισημάνω ότι είχαμε συνολικά κάποιες φιλοδοξίες κάλυψης που θα μπορούσαν να επιτευχθεί με αυτό, καθώς και ε, όσον αφορά τις επιδόσεις αυτών των ευρυζωνικών δικτύων, τις ταχύτερες, ταχύτερες που είχαν ζητηθεί σε αυτή τη συγκεκριμένη πρόταση, Βλέπετε ότι έχουμε προσδώσει και σε ένα βαθμό δυνατότητες ε, όπως υπάρχουν σήμερα στην αγορά και τότε στην προηγμένη τεχνολογία. Και αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται σε αυτό το πρόγραμμα διότι χρειάζεται να έχει πολλαπλασιαστικές ε, επιδράσεις. Αυτό είναι σημαντικό. Δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη κάλυψη, αλλά πρέπει να επιλέξουμε τις υπηρεσίες που θα, τα έργα που θα πολλαπλασιάσουν τα αποτελέσματα και θα προσελκύσουν επενδύσεις που θα έρθουν ως αρρωγή προς τα διευθυντικά ταμεία και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ε, ενώ λοιπόν δεν μιλάμε για υπερβολικά γρήγορο και πάνω από ένα γίγαμπιτ, Μιλάμε για ανάπτυξη εξελιγμένων τεχνολογιών σε αυτά τα έργα και να είναι βασισμένα σε προηγμένα επιχειρηματικά μοντέλα και να υπάρχει δυνατότητα αναπαραγωγής. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι που έχει συμπεριληφθεί σε αυτή την πρόταση. Ένα από τα πράγματα που και εμείς ε, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μας ικανοποιεί είναι ότι έχουμε τόσο σημαντική περικοπή του προπολογισμού. Ωστόσο πιστεύουμε ότι αυτό δεν είναι μήνυμα ότι δεν λαμβάνεται σοβαρά η ψυχική οικονομία. Έχει και μια θετική πλευρά. Αυτή η αρνητική πλευρά του προπολογισμού είναι ότι αποτελεί μια, αποτέλεσε μια ευκαιρία απλοποίησης της πρότασης. Κατά κάποιο τρόπο είναι πολύ πιο απλή, επικεντρώνεται σε προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος, είναι πολύ το σχέδιο και επικεντρώνεται στις προτεραιότητες και στις προτεραιότητες χρηματοδότησης. Σίγουρα θεωρούμε ότι με βάση όλα αυτά δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε σταθερότητα σχεδιασμού. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα, διότι εμείς θέλουμε να προσελκύσουμε και άλλες μορφές χρηματοδότησης αλλά και να μπορούμε να προγραμματίσουμε την κατάργηση διάφορων ψηφιακών υπηρεσιών και να οικοδομήσουμε σιγά σιγά αυτά τα τουβλάκια, όπως είπαμε ψηφιακών υπηρεσιών που έχουν μεγάλη ζήτηση και που έχουν ήδη οριμάσει. Επίσης καθίσταται σαφές ότι εδώ υπάρχει απέτηση όσον αφορά τις υπηρεσίες να γίνουν σοβαρές προσπάθειες ώστε το ενδιαφέρον που εκδηλώνει η αγορά για αυτές τις υπηρεσίες να μεταφραστεί ενδεχομένως σε συγχρηματοδοτήσεις όχι άμεσα, εξαρτάται από τον τύπο υπηρεσίας, αλλά μακροπρόθεσμα ναι. Υπάρχουν λοιπόν ορισμένες υπηρεσίες ορισμένων τύπων όπου μπορεί να φανταστεί κανείς ότι ε, μπορούμε να έχουμε προσδοκίες εμπορικού ενδιαφέροντος αργότερα και που αργότερα θα μπορέσουν να ενταχθούν σε κάποιο είδους συγχρηματοδότηση. Και θέλουμε αυτό να είναι βιώσιμο και πέραν του 2020. Αυτό έχει να κάνει με τη σταθερότητα σχεδιασμού την οποία αναφέρει πολύ σωστά ο κ. Κρότσμαν τώρα. Όσον αφορά το παράρτημα που είναι αρκετά περιγραφικό όσον αφορά του τύπου των αναμενόμενων έργων και η λογική σταδιακή ανάπτυξη. εμείς πιστεύουμε ότι αυτό θα είναι ένα εργαλείο για να αρχίσουμε σε προγραμματικό επίπεδο να οργανώσουμε προσκλήσεις για υποβολή προσφορών για την ανάθεση των συμβάσεων ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν αυτά τα προγράμματα. Το κλειδί σε όλα αυτά θα είναι ότι οι ψηφιακέ υπηρεσίε και τα ευρωζωνικά προγράμματα έχουν το εξή αποτέλεσμα, ότι κινούν το ενδιαφέρον. Είναι σαφέ ότι αυτά τα πράγματα θέλει ο κόσμο και το ξέρουμε και εμεί, αλλιώ δεν θα είχαμε προτείνει αυτόν τον κατάλογο. Δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο να εξηγήσουμε στου πολίτε ότι οι διασυνοριακέ υπηρεσίε όπω το e-health, ή το e-procurement ε, είναι χρήσιμες, αλλά είμαστε ρεαλιστές. Θα χρειαστεί να αποδείξουν την αξία τους στις αγορές αυτές όπου η χρηματοδότηση σπανίζει. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε και μια προσπάθεια προώθησης να προσελκύσουμε χρήση, χρήστες και αυτό αποτελεί κομμάτι του προγραμμάτος ε, αηφορίας και βιωσιμότητας. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτό αποτελεί μια ευκαιρία να υπερασπίσουμε το πόσο λογική είναι αυτή η επένδυση, πώς θα... Αυτές οι ψηφιακές υπηρεσίες ε, συνδέονται με τις εθνικές υποδομές, θα υπάρχουν ε, συνδέσεις με εθνικά κέντρα, όπου κανείς θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε μητρώα ηλεκτρονικής υγείας. Και αυτό είναι ένα πρόσθετο κομμάτι της με το εθνικό επίπεδο, το οποίο θα απαιτούν οι ψηφιακές υπηρεσίε αυτέ σε όλη την Ευρώπη και η χρηματοδότηση κατά την εκτίμησή μα θα μπορέσει να καλύψει μέρο αυτών των συνδέσεων αλλά όχι όλε. Θα χρειαστεί λοιπόν να δημιουργηθεί και ενδιαφέρον σε εθνικό επίπεδο από τις σχετικέ υπηρεσίες ώστε να υλοποιήσουν το μέγιστο αριθμό συνδέσεων στο πλαίσιο του διευρωπαϊκού αυτού πυρήνα που θα υλοποιήσουμε εμείς συνδέσεων. Πρέπει λοιπόν να ζήσουμε με αυτή τη μείωση προπολογισμού. Η πρόταση πιστεύω μπορεί να το αντιμετωπίσει, αλλά χρειάζεται μια αξιόπιστη προσπάθεια με συγκεκριμένε προσπάθειε κατά έργο, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρχει ορίμανση και αηφορία. Ευχαριστούμε για να κλείσουμε. Ο συνάδελφο του Ζενόσκη, παρακαλώ. Eh, Δεν ξέρω τι θα θέλετε να προσθέσω. Στην διάρκεια της συζήτησης ε, των τελευταίων μηνών αποκρισταλώθηκαν πολλά στοιχεία. Φυσικά τώρα αλλάζει η προσέγγιση καθώς γίνονται τόσο μεγάλες περικοπές που ουσιαστικά ένα δέκατο του αρχικού ποσού παραμένει στη διάθεσή μας. Γι' αυτό θα πρέπει να ξεκαθαριστούν και οι όροι, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα πιο στα, στα έργα εκείνα τα οποία είναι πιο πολλά υποσχόμενα. Νομίζω με τόσο περιορισμένους πόρους θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθούν τα έργα που αφορούν την ευρυζενικότητα. Αλλά οι υπηρεσίες αυτές είναι εκείνες που περιγράψαμε. Γι' αυτό λοιπόν θα χρειαστεί ένας νέος ορισμός. Ελπίζω σε αυτή τη συντομευμένη εκδοχή να καταφέρουμε κάτι να πετύχουμε. Θα συνεργαστούμε με τους και εισηγητές, προκειμένου να καταρτήσουμε ένα έγγραφο το οποίο θα μας επιτρέψει να εγκρίναμε το κείμενο στην τελευταία σύνοδο πριν το θερινό διάλειμμα. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα σημεία τα οποία τροποποιήθηκαν σε σχέση με το αρχικό κείμενο και πρέπει να σας πω ότι είμαι αισιόδοξο ότι θα είναι καλή η συνεργασία μας. Ελπίζω να κρατεθούν όλες οι τροπολογίες μέσα στην εβδομάδα και στην περίπτωση αυτή θα διοργανώσω ε, συνάντηση με τους κοιόδες εισηγητές και θα οργανώσουμε τις εργασίες μας ε, μέσα στο χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφος Κράτσμαν ήθελε να κάνει μια άλλη ερώτηση. Όχι, ευχαριστώ πολύ. Η μόνη ερώτηση για την οποία δεν έλαβα απάντηση είναι το πιο ασφαλές διαδίκτυο. Ο κύριο Τίμερς μου έδωσε μια απάντηση, αλλά ίσως να στείλω καλύτερα μια επιτροπή στον Επίτροπο, στην Επιτροπή για να της υπενθυμίσω το ζήτημα αυτό, διότι είναι πολύ ενδιαφέρον ως θέμα και θεωρώ ότι τα ποσά δεν είναι τόσο υψηλά. Μπορούμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμα, πιστεύω. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Υπενθυμίζω ότι η ψηφοφορία στην Ήτρε. Οι τροπολογίες μάλλον θα έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων 19 Ιουνίου και μετά προθεσμίες 25 ε, Ιουνίου το μεσημέρι και 9 Ιουλίου ψηφοφορία στην Ήτρε. Διακόπτε εδώ η συνεδρίαση. Υπενθυμίζω ότι η επόμενη συνεδρίαση θα είναι 19 και 20 Ιουνίου το πρωί και το απόγευμα. Ευχαριστούμε. Καλή δουλειά.